Θα πρέπει πρώτα να κάνουμε το τεστ για να δούμε αν λειτουργεί το μηχάνημα. Αν θέλετε βάλτε τις κάρτες σας, αρχίζει η ε, ψηφοφορία, ψηφίστε ό,τι θέλετε. No, we have to wait. Can everybody vote because δεν ψήφισαν όλοι από ό,τι βλέπω. Μας ε, λείπουν τρεις, δύο τώρα ψήφοι. Δικό σας πρόβλημα είναι έτσι, δεν έχουν ψηφίσει οι δύο. Κάποιοι δεν ψήφισαν. Ας αρχίσουμε λοιπόν την ε, ψηφοφορία. Πρώτα το 8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 αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή 23 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται, 24 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, συμβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, 32 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, 30 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 29 με προφορική τροπολογία. Υπάρχει κανείς που ενίσταται, όχι. Καλά, ψηφίζουμε όπως τροποποιήθηκε, υπέρ, κατά. Εσείς είστε, αλλά είστε κατά. Α, είστε υπέρ, ωραία. Εγκρίνεται λοιπόν. 33, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή. Με ονομαστική ψηφοφορία, ηλεκτρονική δηλαδή, το σχέδιο στο σύνολό του, αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Κλείνει τώρα. Εγκρίνεται με 35 υπέρ, μία κατά. Συγχαρητήρια. Το 9. Γνωμοδότηση Μιράντα για τις μικρής κλίμακας αλίες και την ε, μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 5. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται αυτή. Τροπολογία 6 με προφορική τροπολογία. Υπάρχει κάποια ένσταση. Όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν όσο τροποποιήθη υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 8 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή. 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία τώρα για το σχέδιο γνωμοδοτήσεως, στο σύνολό του, αρχίζει. Πέρας. Πάλι 35 προς 1 εγκρίνεται και συγχαρητήρια την Μιράντα. Είναι και η πρώτη σας ψηφοφορία, έτσι δεν είναι. Ακολουθεί του Όλτριχ Βλάσακ. Συγγνώμη. Μου επιτρέπετε να λάβω το λόγο. Είναι η πρώτη μου ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με μεγάλη μου χαρά. Και ευχαριστώ και για, τα, και για τις συμβαστικές. Ωραία. Το 10. Όλτριχ Φλάσακ. Το σχέδιο γνωμοδοτήσεω για την ελκυστικότητα επενδύσεων στην Ευρώπη. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Τώρα. Ακολουθεί συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται και αυτή. 18. 18 ε, επαναλαμβάνω υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Μπορούμε όμως και να το επαληθεύσουμε αν θέλετε. Ας επαληθεύσουμε. Την 18. Νομίζω ότι είναι σαφώς κατά, αλλά ας επαληθεύσουμε. Ίσως και πηγαίνουμε και πολύ γρήγορα. Λοιπόν, απερίφθη. Τώρα, 19 υπέρ κατά. Εδώ πραγματικά δεν μπορώ να πω. Ας κάνουμε παλήθευση λοιπόν για τη 19. Ψηφίζουμε τη 19 λοιπόν, αρχίζει η ψηφοφορία. Ναι, έχει αρχίσει η ψηφοφορία. Την 19. 19. Η 18 εγκρίθηκε προηγουμένω. Ή μάλλον απερίφθη, λέει ο πρόεδρο. Απερίφθη διορθώνει ο πρόεδρος. Πέρας τώρα τη ψήφου. Εγκρίνεται με διαφορά δύο ψήφων. Η 20 υπέρ. Κατά. Πάλι πρέπει να επαληθεύσουμε. Δεν είναι σαφές. Για την 20 λοιπόν. Αρχίζει. Πέρας. 20 υπέρ 16 κατά εγκρίνεται. 21 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται νομίζω και αυτή. Νομίζω είναι και ο ίδιος συσχετισμός των δυνάμεων. Πού πηγαίνουμε τώρα. 24. Προπολογία 24. Υπέρ. 24 λοιπόν, εντάξει. Είπε; Καθαρά παρακαλώ, καθαρά τα χέρια. Κατά. Καλά, θα επαληθεύσουμε. 24. Αρχίζει η ψηφοφορία. Απορρίπτεται 24. 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται χρειάζεται παρήθευση, όχι 22 22 κάνουμε παρήθευση. αρχίζει η ψηφοφορία πέρας 21 κατά 18 υπέρ. Άρα απορρίπτεται. 23 υπέρ. Κατά. Η ίδια δύσκολη κατάσταση. Ας επαληθεύσουμε πάλι για την 23 λοιπόν. Πέρας. Εγκρίνεται με διαφορά τριών ψήφων 25. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή 28 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι αυτή απορρίπτεται αλλά ας επαληθεύσουμε 28 αρχίζει πέρας Απερίφθη με τρεις ψηφοδιαφόρα. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Αυτή απορρίπτεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας επαληθεύσουμε την 31. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ποτέ δεν είχαμε τέτοια διέρεση στη μέση. Εσείς πάντοτε καταψηφίζετε. Τέλος πάντων, τώρα τελείωσε και απερίφθη με τρεις ψήφους διαφορά. 29. Κωνσταντσε, τι θα δείξετε εσείς. Τι νόημα θα κάνετε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση και εδώ. Είναι πολύ κοντά η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε. Πάμε στην 32. Ψηφί υπέρ στις 32. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές Νομίζω ότι αυτή εγκρίνεται, αλλά ας, το επαληθεύσουμε. Πέρας και εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Ας, ας επαληθεύσουμε όμως. Συμβαστική 3. Πέρας. Εγκρίθηκε λοιπόν. Άρα εκπίπτουν οι υπόλοιπε. Πάμε στη 43. Υπέρ. 43 παρακαλώ. Καθαρά τα χέρια. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. Ακόμα και το Λαϊκό Κόμμα είναι διαιρεμένο ή σηκώνετε τα χέρια σας με καθυστέρηση. Όχι εσείς ειδικά, οι συνάδελφοι γενικά. 22 ναι. υπέρ, 17 κατά. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές. Πάλι δεν είμαι βέβαια. Ας επαληθεύσουμε τη 44. Είσαστε πάρα πολύ κοντά τα δύο στρατόπεδα. Ένα ή μία δεν ψήφισε. Πάντω έχει εγκριθεί με τέσσερις ψήφους διαφορά. Συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τώρα ακολουθεί η 49. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 52. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 53. Υπέρ. Κατά. αποχέ. εγκρίνεται. 54 υπέρ. Κατά. Ας επαληθεύσουμε την 54. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίθηκε πράγματι, σαφώς μάλιστα. 55 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. 55. Αρχίζει. πέρασε Και εγκρίθηκε. 25 19 κατά. 56 υπέρ. Κατά. Και εδώ χρειάζεται παρήθευση. 56 λοιπόν αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρασε, Εγκρίθηκε. 57 υπέρ κατά. Επαλήθευση, λυπούμε, αλλά δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Πέρας. Εγκρίνεται με 20 προς 18. 58 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 59 υπέρ, κατά, Επαλήθευση. Αρχίζει η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίφθηκε αυτή. Τώρα, θέτω σε ψηφοφορία το σύνολο της ε, γνωμοδοτήσεως με ηλεκτρονική ψηφοφορία που έχει αρχίσει. Κάποιος, ένα, ένα πρόσωπο δεν έχει ψηφίσει. Αν θέλετε όμως μπορούμε να κλείσουμε την ψηφοφορία. Εγκρίθηκε λοιπόν 32 προς 4 και δύο Τελειώσαμε την ψηφοφορία αυτή. Τώρα ο Βίκτορ Ποστινάρου, αλλά η Κομισιόν δεν είναι ακόμα παρούσα. Λυπούμε κύριε Ποστινάρου, η Κομισιόν θα έρθει όμως φαντάζομαι. Μάλλον εγώ ήθελα ο εκπρόσωπος της Επιτροπής της Κομισιόν να ολοκληρώσει τα σχόλια. Μήπως περιμένει ο άνθρωπος έξω. Δεν είναι λοιπόν παρούσα ακόμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε θα ξεκινήσουμε με το καινούριο σημείο. in κοιτάξτε, θα έρθει σε πέντε λεπτά. Αν ξεκινήσουμε ένα άλλο θέμα θα πρέπει να περιμένει μετά πάλι ώσπου να το τελειώσουμε. Ε, το θέμα είναι να μην δημιουργήσουμε μια κάποια σύγχυση. Αν θέλετε μπορούμε να περιμένουμε. The bus is here. It's your report. If you want to wait five minutes, we can wait. Five minutes is. is better to Lambert prefers to have Victor speaking or what? Θέλετε να μιλήσει ο Victor λοιπόν ή όχι. Α, θέλετε διακοπή, διακοπή λοιπόν για πέντε λεπτά. Τότε να περιμένουμε πέντε λεπτά. Γιατί αλλιώς θα δημιουργηθεί μια σύγχυση. Because they are very far and they are coming. They are coming. I think they are, they are in the building already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 One minute late or two minutes late? No, no, one minute. One minute. <laughs> uh, dear, dear Nicholas, dear director, we just give you 10 seconds to... Σας δίνουμε 10 δευτερόλεπτα να βγάλετε τα χαρτιά σας. Όπως είπαμε μπορείτε να συνεχίσετε τα σχόλιά σας για τη συζήτηση για το γενικό κανονισμό και μετά θα ακούσουμε τους συζητητές και μετά θα δώσω το λόγο στον Βικτόρ Μποστινάρο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Υπάρχουν ορισμένα θέματα σε εκκρεμότητα, όχι πάρα πολλά. Θα ήθελα να συμπληρώσω λοιπόν την παρέμβασή μου σήμερα το πρωί. για τη συζήτηση την πρωινή την οποία παρακολούθησα με πολύ ενδιαφέρον. Σχετικά με το αποθεματικό επιδόσεων η ανησυχία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι αν καταργήσουμε το άρθρο 20 στο σύνολό του, αν το διαγράψουμε, υπάρχει ένας κίνδυνος να πετάξουμε το μωρό μαζί με το νερό του μπάνιο. δηλαδή τι εννοούμε. Λόγω της κατάργησης όχι μόνο του ιδίου του αποθεματικού αλλά και των προβλέψεων που οδηγούν στην διακοπή και την διόρθωση ε, κάποιων στόχων εφόσον έχει υπάρξει αποτυχία επίτευξης των στόχων αυτών. Σε αυτή την περίπτωση, την περίπτωση αποτυχίας, ο μηχανισμός επιδόσεων είναι κάτι το οποίο δεν είναι πλέον κατάλληλο και παρόλα αυτά το πλαίσιο του μηχανισμού υπολογισμού των επιδόσεων είναι κάτι το οποίο εμείς θα θέλαμε να συγκεντρώσει την προσοχή όλων. Πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο και γι' αυτό πιστεύουμε ότι και ε, αυτό το, αυτή η πρόταση, η, το αποθεματικό επιδόσεων, η απόθεμα επιδόσεων, είναι κάτι το οποίο δεν θα είναι υποχρεωτικά ιδιαίτερα βαρύ γραφειοκρατικά και θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο. Τώρα για τη μακροοικονομική αιρεσιμότητα, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχει συζητηθεί επανειλημμένα στην Επιτροπή σας. Αυτό που πρέπει να πω εδώ είναι ότι Εάν πράγματι θέλουμε να έχουμε μια πολιτική η οποία να βασίζεται στην ανάπτυξη και στην οικονομική ανάπτυξη και στην ανάπτυξη των οικονομικών ρυθμών, τότε δεν πρέπει να αποκλείσουμε τη διασύνδεση της διαδικασίας αυτής με την ευρύτερη διακυβέρνηση της οικονομίας. Γι' αυτό θεωρούμε ότι οι προβλέψεις για τη μακροοικονομική αιρεσιμότητα είναι αναπόσπαστο κομμάτι του συνολικού πακέτου που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ίσως σε αυτό το πλαίσιο να υπογραμμίσω ότι η αναλογικότητα την οποία θέσατε είναι σε εισαγωγικά εντυχισμένη στις προτάσεις μας, στις προβλέψεις μας και μπορεί να επηρεάσει πλήρως και ισότιμα όλα τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να μην υπάρχουν μη ομαλές και στρεβλές συνέπειες της εφαρμογής των προγραμμάτων. Τέλος. να φτάσω πάλι στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο. Εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, παραδίδει αυτά που είχε υποσχεθεί ότι θα παραδώσει στα πλαίσια του κειμένου εργασίας το οποίο περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία τα οποία θα περιλαμβάνονται, θα μέσα στην κατεξουσιοδότηση πράξη την οποία εμείς προτείνουμε σχετικά με τους τρόπους με τον οποίο αλληλοεπηρεάζονται τα πέντε ταμεία με άλλους τομείς και άλλα προγράμματα όπως και το πρόγραμμα το στρατηγικό Horizon 2020. Πρέπει λοιπόν και δίδονται κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για την συγκέντρωση την προσοχ... της προσοχής μας σε θεματολογικές εξελίξεις και την περιφερειακή διάσταση και το πώς αυτό μπορούμε να τα διασυνδέσουμε, πώς αυτά μπορούμε να τα διασυνδέσουμε. Και επίσης ε, συνδέουμε την ε, προοπτική αυτή και με το λεγόμενο ευρωπαϊκό εξάμεινο. Λοιπόν, αυτά προσφέρει το έγγραφο όπως είπε και ο κύριος Όλμπρεχτ, δεν είναι ένα νομοθετικό κείμενο, δεν σκοπεύαμε να παρουσιάσουμε ένα νομοθετικό κείμενο, ένα όμως επεξηγηματικό κείμενο παρουσιάζουμε, το οποίο να περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία. Δεν είχαμε τη δυνατότητα να το παρουσιάσουμε στην Επιτροπή σας ακόμα. Είχαμε την ευκαιρία να την την πρότασή μας στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου και να συλλέξουμε και τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνονται τα κράτη-μέλη σε αυτές τις προτάσεις. Και γι' αυτό ήταν πολύ καλή η ευκαιρία που μας δόθηκε να δούμε και τις αντιδράσεις από την παρουσίαση που κάναμε και σε εσάς. Εμείς ε, πιστεύουμε ότι πρέπει να ασχοληθούμε με την ουσία, με το περιεχόμενο της πρότασης και μετά να βρούμε τη σωστή διαδικασία για να δημιουργήσουμε τελικά ένα νομοθετικό κείμενο. Γνώμη μας είναι ότι αφού λάβαμε το feedback αυτό από τα δύο όργανα, από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, που συνομοθετούν, τότε θα δούμε και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς θα προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο επί τη βάση των ε, ενδείξεων των δύο άλλων οργάνων. Πάντως αυτές είναι οι βασικές μας προτάσεις, πρόκειται για μια αρχική πρόταση, μια πρόταση σε αρχικό στάδιο εννοώ και από εδώ θα θέλαμε να προχωρήσουμε έτσι ώστε να μειώσουμε τους ε, κινδύνους που μπορεί να παρουσιαστούν για να έχουμε κάτι το οποίο να είναι εφαρμόσιμο στα προγράμματα τα επιμέρους, τα επιμέρους μία και να αποφύγουμε ένα διοικητικό αδιέξοδο το οποίο θα υπονομεύσει τους κοινού μας στόχους. Τέλος, να ανταποκριθώ λίγο και στα σχόλια της κυρίας Κρέλ για, τις, για τη μελλοντική συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να σας διαβεβαιώσω ότι εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε να στηρίζουμε από πλευράς επιτροπές, επιτροπής τις προσπάθειες των εισηγητών και τις προσπάθειες της Επιτροπής σας. Θεωρούμε ότι κάνετε επικοδομητικά πράγματα, θεωρούμε ότι έχουμε αρκετές κοινέ θέσεις και θα καταλήξουμε από κοινού σε ένα νομοθετικό κείμενο που να σέβεται τις βασικές αρχές αλλά να παρέχει όμως και το απαιτούμενο, το σωστό νομοθετικό πλαίσιο έτσι ώστε να μπορέσουμε να προσελκύσουμε τις επενδύσεις που χρειάζεται και να πετύχουμε τους στόχους μας. Έχουμε διαφορετικές απόψεις σε ορισμένους τομείς. Σε κάποιους από αυτούς εμένουμε σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί θεωρούμε ότι το διακύβευμα είναι σοβαρό αλλά θεωρούμε επίσης από τις επαφές που είχαμε ότι τα σχόλια είναι επικοδομητικά και οι διαφωνίες είναι περιορισμένες. Σας ευχαριστώ. Φαντάζομαι ότι και οι συγητές θα ήθελαν να λάβουν το λόγο για σχόλια. Ποιος πρώτος, ο Λάμπερτ. Μιλήσετε για στόκευση. Ωραία. Η ίδια η αρχιτεκτονική πάντως της πρότασης κρατάει σταθερό το σύστημα για την ολοκληρωμένη προσέγγιση, θα υπάρξει ευρεία κάλυψη. Έτσι θα εξασφαλιστούν και τα αποτελέσματα. Όλα αυτά τα επιμέρους σημεία είναι πολύ σημαντικό και για το στρατηγικό πλαίσιο, αλλά και γενικώ συμφωνούμε με τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. και νομίζω ότι θα πρέπει να λιλιποστηριχθούμε στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Γιατί δεν είναι σαφές ακόμη τι θέση θα κρατήσει το Συμβούλιο. Πάντως, ελπίζω μέχρι στιγμή οι συνάδελφοι να έριξαν μια ματιά στις τροπολογίες για να συμβάλλουν και αυτοί με τις προτάσεις τους στον εμπλουτισμό της συζήτησης πολλές τροπολογίες θα είναι παρόμοιες, οπότε δεν περιμένουμε ιδιαίτερες εκπλήξεις. Τώρα, όπως είπαν και ο κύριος Γκοντμάνης ε, και άλλοι συνάδελφοι, σε αυτή τη φάση δεν ασχοληθήκαμε με συγκεκριμένα νούμερα. Και η κρατούσα γνώμη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι επιφυλακτική ως προς τη μνήμα συγκεκριμένων αριθμών σε αυτή τη φάση. Πάντως στο δεύτερο, στη δεύτερη δόση των τροπολογιών, στο δεύτερο τμήμα ε, και σε επίπεδο έκθεσης Γκαρίγκα θα κάνουμε συγκεκριμένες ε, προτάσεις. Πάντως το θέμα της προσέγγισης θα το αφήσουμε ανοιχτό, αλλά θα αναφέρουμε την ε, υποστήριξή μας στη θέση της έκθεσης Γκαρίγκα. Περιμένουμε φυσικά τους υπολογισμούς του κυρίου Γκοντμάνης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο για τα επόμενα βήματα. Θα δούμε αν είναι ισορροπημένες οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Φυσικά για το κάπινγκ, για το καθορισμό αναδοτών ορίων, ο καθένας μπορεί να έχει τη γνώμη του. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα για όλους και θα ενταχθεί στη συζήτηση για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Πάντως πρέπει να διαμορφώσουμε και τη δική μας γνώμη για το καθορισμό ανά τον για το κάπινγκ. Πάντως περιμένουμε, παραλαμβάνουμε ενδιαφέρον τα στοιχεία, τους αριθμούς που προκύπτουν από τους υπολογισμούς του κ. Κοντμάνης. αναφέρθηκαν κάποιες αμφιβολίες για την προσέγγιση. Αλλά προς το παρόν είμαστε διαλλακτικοί και προσπαθούμε να υιοθετήσουμε μια νομική εμπειρία για ένα κείμενο που θα πρέπει να περιλαμβάνει στο διατακτικό αυτό που αναφέρεται στο παράρτημα. Είπαμε να μπει στο παράρτημα αυτό φαίνεται προέκυψε και από τη σημερινή συζήτηση, να γίνει προ το παρόν τώρα και να το συζητήσουμε αργότερα. Πάντω, αυτό που σημείωσα από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι θα συνεχιστεί η συζήτηση και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πάντως η θέση του Κοινοβουλίου είναι σαφή. Δεν υπάρχει αδιέξοδο. Γιατί είμαστε συνεπεί με αυτά που είχαμε πει και στο παρελθόν. Και όπως είπατε, είμαστε και συνομοθέτες εδώ. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εταιρική σχέση, εταιρικότητα, προσπαθήσαμε να αναφέρουμε τις τοπικές και περιφερειακές ε, αρχές πρώτες και μετά σε εταιρική σχέση με τα υπόλοιπα. Προσοχή λοιπόν ε, να ξαναδιαβάσουμε το κείμενο και είπε η κυρία Σρέντερ ότι αποκλείσαμε του, την, τις τοπικές αρχές. Όχι, φυσικά και όχι μάλλον παρεξήγηση δημιουργήθηκε. Ουδέποτε δεν αποκλείσαμε τις τοπικές περιφερειακέ αρχέ. αρχές. Κώδικα συμπεριφορά. Από ό,τι φαίνεται έχει σταλεί, αλλά δεν τον κοίταξα ακόμη. Θα πρέπει να τον εξετάσουμε ενδελεχώ. Και φυσικά και εδώ χρειαζόμαστε ισορροπημένη προσέγγιση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη σχέση με τους ειδικού κανόνες για τα ταμεία. Ε, ισχύει για το ΕΚΤΑ και το ΦΕΝΤΕΡ. Καλό θα ήταν να πούμε όπου δει, όπως ζήτησε ο κύριος Όλμπριχτ, μια διευκρίνηση δηλαδή. σε πολλές περιπτώσεις προβληματιστήκαμε για την ερμηνεία ε, του κειμένου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 38.1 για παράδειγμα αναφέρεται ο, στόχο, στόχος, aim, στοχεύει. Μετά αντικαταστάθηκε από θεματικούς ειδικού στόχους. Νομίζω ότι αυτό ευθυγραμμίζεται με διατύπωση άλλων σημείων του κανονισμού. Σε πολλά σημεία διευκρινίσαμε το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πάντως θα δούμε ποια είναι η προστιθέμενη αξία ως προς τη συμπληρωματικότητα των ταμείων στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο των ταμείων και θα περιορίσουμε το εργαλείο αυτό εκεί που χρειάζεται, εκεί που έχει προστιθεμένη αξία και θα περιοριστούμε φυσικά και στο νομικό κείμενο. Ευχαριστώ θερμά τους συναδελφούς για τις προτάσεις τους. Θα εξετάσουμε το κείμενο τις επόμενες μέρες και θα το συμπληρώσουμε και με άλλες τροπολογίες. Πάντως, έχω καλό προέστημα για την προθυμία και των μελών της Επιτροπής και των ε, ειδικών εισηγητών. Ε, έχω καλό προέστημα ότι θα προλάβουμε να ολοκληρώσουμε την ψηφοφορία πριν το καλοκαίρι είναι εφικτό κάτι τέτοιο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί έχουμε πολλά υπουργικά συμβούλια που αναμένονται να γίνουν και ίσως προκύψουν κάποιες αμφιβολίες, αλλά αυτό είναι θέμα του Συμβουλίου, όχι του Κοινοβουλίου. Το πρωί η Κωνσταντζα μια χαρά τα πήγες, σε ακούμε και τώρα. Σύμφωνοι. Στα αγγλικά η κυρία Κρέλ. Έχω λίγα σχόλια. Τέθηκε το θέμα της έναρξης του επιχειρησιακού προγράμματος τρεις μήνες μετά από την σύνταξη της εταιρική σύμβασης. Δεν είναι ακριβώς έτσι μέχρι ε, να περάσουν τρεις μήνες έτσι. Επικύρει από την κατάσταση την οποία βρίσκεται το κράτος μέλος. Εάν όλα είναι έτοιμα μπορεί να αρχίσει η συνάντηση και με το επιχειρησιακό πρόγραμμα και με την εταιρική σύμβαση ταυτόχρονα ή πάντως μέσα στο διάστημα των τριών μηνών αν χρειάζεται περισσότερη επεξεργασία το operational program. Αυτή είναι μια χρήσιμη, ένα χρήσιμο στοιχείο ευκαμψίας. Έγινε και μια ερώτηση νομίζω από την κυρία Μανέσκου ανάμεσα, μια διάκριση ανάμεσα στο must και στο shall. Αυτά βέβαια είναι η νομική γλώσσα. Δεν, δεν έχουμε εμεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε τις ε, λέξεις στα αγγλικά must ή have to. Το, το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι shall. Αυτή είναι η εξήγηση, αυτή είναι η απάντηση στην ερώτησή σας. Ένα άλλο που τέθηκε ήταν για το χρονοδιάγραμμα που χρησιμοποιούμε για τη δυνατότητα στήριξης μιας περιφέρειας. Το πιο επίκαιρο που έχουμε, όπως γνωρίζετε, είναι από τα έτη 2007, 2008 και 9. Και αν δεν είμαστε έτοιμοι μέχρι τον Μάρτιο του χρόνου, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τα έτη 2008, 9 και 10. Για ορισμένες περιπτώσεις αυτό ισχύει, για άλλες όχι, αλλά πάλι δεν είναι δική μας απόφαση αυτή. Εμείς πάντως βασιζόμαστε στα πιο πρόσφατα νούμερα που διαθέτουμε. Έρχομαι ξανά στην ερώτηση του Γιάννη για τους εξειδικευμένους κανόνες. Όπως είπε ο Λάμπερτ Βανίστερ Ρο, είπε ότι ο στόχος δεν έχει καθοριστεί ακόμα. Στο δε άρθρο 87 1 β και ε, συγγνώμη, 2 β και ε, έχετε τους ειδικού στόχους για κάθε άξονα προτεραιότητας. Σε συσχετισμό δηλαδή με αυτούς τους ειδικού κανόνες και γι' αυτό είπαμε ότι πρέπει, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και ειδικού στόχους. Εν τέλει θα πρέπει να το ελέγξουμε, αλλά αυτή είναι η ιδέα που κρύβεται πίσω από αυτό. Επίσης έγινε μια ερώτηση για τα κριτήρια και τους δείκτες για την λίστα για λειτουργικές αστικές περιοχές. Αυτό το συζητήσαμε και με τον εισηγητή και με τον Γιάν για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Ανάπτυξης, γιατί η πρότασή του ήταν να υπάρχει ε, μια τέτοια ε, λίστα δικτών για να δείχνει τι είναι μια λειτουργική αστική περιοχή. Μπορεί να είναι μια Μητρόπολη, μπορεί να είναι ένα αστικό κέντρο, μπορεί να είναι και η περιφέρεια ενός αστικού κέντρου ή ένα τμήμα της πόλης, αλλά χρειαζόμαστε κάποια κριτήρια αυτό λοιπόν είναι το κείμενο που συντάξαμε και τα υπόλοιπα θα μας έλθουν από τον Γιάννη και την έκθεση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Αυτά ήταν νομίζω τα ανοιχτά ερωτήματα που είχα σημειώσει. Πάντως η δική μου εντύπωση ήταν ότι η συζήτηση του σημερινού πρωινού ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη για, τους, για μας τους συζητητές, διότι έχουμε ήδη κατά νου τις τροπολογίες που θα υποβάλουμε τέλη Μαΐου και έχω την εντύπωση ότι αυτά τα ζητήματα που θέσατε στη συζήτηση του σημερινού πρωινού, πολλές από τις ιδέες αυτές ήδη έχουν μπει σιγά σιγά στις τροπολογίες της επόμενης δόσης και νομίζω ότι έχουμε τη βάση για να καταλήξουμε σε μια θέση στην Επιτροπή που να υποστηριχθεί από τη μεγάλη πλειοψηφία των μελών. Βέβαια, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να ικανοποιήσουμε 100% όλους, αλλά ε, να μπορέσουμε να εξεύρουμε μια στρατηγική που να μας επιτρέψει να προωθήσουμε την πολιτική συνοχή στα επόμενα χρόνια. Νομίζω ότι με τον τρόπο που περιέγραψα θα πετύχουμε σημαντική πλειοψηφία που να μπορεί να ακολουθήσει αυτό το ερυθρό νήμα το οποίο θα οδηγεί προς το μέλλον. Νομίζω ότι βοήθησε πολύ λοιπόν η συζήτηση αυτή. και πολύ ενδιαφέρον ενδιαφέρουσα συζήτηση για το Code of Contact. Είδα και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σήμερα το πρωί. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Και θα δούμε τώρα πώς θα προχωρήσουμε. Σας ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστώ. Οπότε μπορούμε να ολοκληρώσουμε το σημείο 4 της ημερήσης διάταξης και να πάμε στο 11, την έκθεση Μποστινάρου για το Ταμείο Συνοχής. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Έχουμε μέχρι στιγμής μόνο την αγγλική εκδοχή του κειμένου για το Ταμείο Συνοχής. Το κείμενο αυτό αντανακλά μακροσκελή συζητήσεις που είχαμε στην Επιτροπή, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο και εγώ ως με τους και οδησηγητές ε, επίσης ε, συζητήσαμε το θέμα. Είχαμε πολλές διαβουλεύσεις με, με κυβερνητικές οργανώσεις, με εκπροσώπους των κυβερνήσεων, με εξαίρεση τη ρουμανική κυβέρνηση, με ε, επιχειρηματίες και εκπροσώπους των περιφερειών. Όλα αυτά, ο καρπός όλων αυτών των διαβουλεύσεων περιλαμβάνεται στο σχέδιο έκθεσης. Όπως βλέπετε, δύο είναι οι βασικές τροπολογίες στην έκθεσή μου. Η πρώτη αφορά τη στήριξη του Ταμείου Συνοχής για, θέματα ενεργειακής για σχέδια ενεργειακής αποδοτικότητας και χρήση ενώσιμων πηγών ενέργειας στον τομέα της στέγασης και ε, η στήριξη των ε, ε, εργοστασίων συμπαραγωγής ενέργειας θερμότητας ε, για την ε, θέρμανση και ψήξη της πόλης. Επίσης, ε, προτεραιότητες επενδυτικές. Ο λόγος για τον οποίο κατέθεσα τις τροπολογίες είναι γιατί θέλουμε να περιλάβουμε την ενεργειακή αποδοτικότητα σε θέματα στέγης για την επιλεξιμότητα των κονδυλίων του Ταμείου Συνοχής. Έτσι θα βελτιώσουμε την ενεργειακή αποδοτικότητα και θα υλοποιήσουμε τους στόχους της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για το 2020. Γνωρίζουμε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από άλλες πηγές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προσπαθήσει να τηρήσει τους στόχους της του 2020 για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Και αν συνεχίσουμε την παρούσα τάση, θα καταφέρουμε μόνο λίγο κάτω από το 10% να επιτύχουμε το στόχο, ενώ αν αν αυξήσουμε την ενεργειακή μας αποδοτικότητα μπορούμε να φτάσουμε και σε τουλάχιστον 20% ποσοστό. Έτσι θα κάνουμε πιο φιλοπεριβαλλοντική την οικονομία μας και θα υλοποιήσουμε τους στόχους της στρατηγικής του 2020. Πάντως, οι στόχοι Ευρώπη 2020 δεν είναι ο μόνος λόγος για να στηρίξουμε τέτοιου είδους σχέδια θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι θα αποτελέσουν έναυσμα για την πράσινη οικονομία και για πραγματικά φιλοπεριβαλλοντικές θέσεις απασχόλησης και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης θα, μειωθούν οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, άλλο σημαντικό στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα γίνουν και σημαντικές οικονομίες ε, στα νοικοκυριά που θα βλέπουν ε, τους λογαριασμούς ε, της ενέργειας να μειώνονται γιατί μέχρι στιγμής ε, οι λογαριασμοί της ενέργειας είναι υπαρθμόν ένα εχθρό σε όλες τις χώρες. Επίσης υπάρχει το θέμα της ε, ασφάλειας του ενεργειακού ενεφοδιασμού της Ένωσης. Ο τομέας ε, ο οικοδομικός αντιπροσωπεύει το 40% και το τονίζω το 40% του, της συνολικής πανευρωπαϊκής χρήσης ενέργειας και 36% των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, κάτι που δείχνει ότι έχει τεράστιο αποτέλεσμα ε, η στήριξη του οικοδομικού τομέα στην υλοποίηση των στόχων. Και μάλιστα η συνέργεια μεταξύ Ταμείου Συνοχής και ΕΤΠΑ, Ταμείου Περιφερειακή Ανάπτυξης, θα, θα προωθήσει τις ε, επενδύσεις ε, στον, στον ενεργειακό τομέα, στον οικοδομικό κλάδο και φυσικά θα καλύψει τις ανισότητες μεταξύ των περιοχών λόγω των διαφορετικών κριτήριων επιλεξιμότητας. Επίσης, το Ταμείο Συνεχής θέλει να, να στηρίξει ε, αποτελεσματικά εργοστάσια συμπαραγωγής ενέργειας θερμότητας ε, και θέλουμε να μιλούμε όχι μόνο για συμπαραγωγή, δηλαδή θερμότητα και ηλεκτρισμό ή θερμότητα και ψήξη. Στη Γερμανία, την Αυστρία, τη Βιέννη, ήδη έχουμε εργοστάσια και σχέδια για την τελευταία γενιά της ε, συμπαραγωγής και μπορεί να γίνει και μια μετατροπή από τα ορυκτά καύσιμα στην παραγωγή ενέργειας με ανανεώσιμες πηγές και αυτό είναι το μέλλον. Θέλουμε αυτό το παρθένο σχετικά έδαφος, το εξερεύνητο, να το εξερευνήσουμε περαιτέρω. Είναι σημαντικό για τις μελλοντικέ εξελίξεις. Τώρα, έχουμε εδώ εργοστάσια που είναι αποτελεσματικά και αποδοτικά εξαιτία ε, της σχέσης που έχουμε μεταξύ ε, κατανάλωσης καυσίμων, επίπεδου καυσαερίων και ωφέλειας για τις κοινότητες και για τον τομέα στέγασης γενικώ. Τα εργοστάσια συμπαραγωγή στην θερμότητα ψήξη των πόλεων στηρίζονται από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής και έχουν μεγάλη σημασία για τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει λοιπόν να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Συνοχή, όχι επειδή ε, είναι συχνά να, έχουν, να υπάρχουν τέτοια εργοστάσια, αλλά επιτρέπουν σημαντικέ οικονομίε ε, και ω προ τη ρήπαση, αλλά και ω προ τι δαπάνε τι ενεργειακέ των οικοκυριών. Σε πολλέ χώρες έχουμε περάσει από ε, συλλογικά συστήματα σε ατομικά συστήματα, που είναι πιο δαπανηρά, πιο ενεργειοβόρα και εκπέμπουν περισσότερες εκπομπές διεξιδίου, του άνθρακα. Ούτε ωφελούν ιδιαίτερα κοινότητα, την κοινότητα, την κοινωνία, τα κράτη-μέλη, ούτε θα μας επιτρέψουν να υλοποιήσουμε του στόχου του 2020. Οι επενδύσει λοιπόν στον τομέα αυτό θα πρέπει να συνοδεύονται από κίνητρα. Και παραλαμβάνω, εργοστάσια υψηλής αποτελεσματικότητας, γιατί χρησιμοποιούν καλύτερες τεχνολογίες, αποτελεσματικές, φιλικές προς το περιβάλλον, χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πόνες ενέργειας και άρα εξασφαλίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια. Επίσης θα βοηθήσουν τη μείωση των ενεργειακών δαπανών των πολιτών και θα αποφευθεί και η χρήση ιδιωτικών συσκευών, ατομικών ε, συσκευών. Πολύ σημαντικά στοιχεία είναι η συμβολή του Ταμείου Συνοχής ε, στην ε, ανάπτυξη των πόλεων. Για πολλούς συναδέλφους η ανάπτυξη των πόλεων είναι νευραλγικός ε, παράγοντας για τον εξυγχρονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια απτή συμβολή και αποτελεσματική και επίσης θα μας επιτρέψει να υλοποιήσουμε και θεματικούς στόχους Λαμβάνοντα και πάλι υπόψη τη συμβολή του Ταμείου συνοχή. Και όταν έχουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση τον παραγωγό, τον μεταφορέα της ενέργειας, τη ηλεκτρισμό, θέρμανση, ψήξη και χρησιμοποιούμε αυτά τα τελέσματα της παραγωγής με σύγχρονα κτίρια, με οικονομία ενέργειας, θα έχουμε τεράστια ωφέλη και για την κοινωνία και για τα κράτη-μέλη. Σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες. Οι τροπολογίες αυτές είναι η αφετηρία. Θέλουμε καλύτερο ορισμό, αποφυγή των παρεξηγήσεων και να βρούμε τον καλύτερο τρόπο για την ε, πολιτική συνοχή του μέλλοντος. Επίσης, ε, αναφέρονται οι υποδομές που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής και η πρόσβαση των ε, ατόμων με αναπηρίες ή με περιορισμένη κινητικότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ε, κυρώσει την σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ανθρώπων, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ευθυγραμμιζόμαστε με τη σύμβαση αυτή του ΟΗΕ Επίσης, οι τροπολογίες που υπέβαλα ευθυγραμμίζονται και με τις υπόλοιπες ε, πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μιλούν για την ανάγκη εξασφάλισης ε, της ε, πρόσβασης των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες στις διάφορες υποδομές. Έχουμε νέα αιτιολογική σκέψη για διευκρίνηση της σχέσης μεταξύ Ταμείου συνοχή και της αρχή ορυπαίνων πληρώνει. Με διαβεβαίωσαν ότι Πολύ σύντομα ο Επίτροπος Ποτότσνικ θα υποβάλει το σχέδιο οδηγίας για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Την περιμένω λοιπόν, γιατί ίσως προταθούν κάποιες αλλαγές στη μελέτη επιπτώσεων του στρατηγικού περιβάλλοντος, ώστε να αποφύγουμε διασπάθηση των κονδυλίων ε, του Ταμείου Συνοχής για περιπτώσεις που ο δεν πληρώνει. Επίσης, η του Natura 2000 ως ε, μηχανισμού προστασίας της βιοπικιλότητας. Κάτι που παραλυπόταν από το σχέδιο κανονισμού, ενώ είναι πολύ σημαντικό για την υλοποίηση των στόχων μας. Επίσης, η περίληψη της υπαίθρου ε, είναι πολύ σημαντικό παράγοντας, γιατί ορισμένα προγράμματα και σχέδια δεν μιλά μόνο για αστικές περιοχές και προάστια, αλλά και περιοχές γύρω από τις πόλεις. Θα πρέπει λοιπόν να υιοθετήσουμε και εδώ ολοκληρωμένη προσέγγιση. Επίσης, θέλουμε να ενθαρρύνουμε την κινητικότητα των πολιτών. Καλύτερα να μιλάμε για τέτοια κινητικότητα παρά για κινητικότητα της πόλης. Επίσης, έτσι θα περιορίσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και θα κάνουμε πιο φιλοπεριβαλλοντικές τις συγκοινωνίες και τα δημόσια μέσα μεταφοράς. Πάντως, πιστεύω ακράδαντα ότι θα συνεχιστεί η αγαστή συνεργασία που είχαμε με τους κοιόδης ηγητές, τους οποίους ευχαριστώ θερμά για τη συνεισφορά τους και για την προθυμία τους για στενή συνεργασία. Πιστεύω ότι θα συνεχιστεί αυτή, αυτό το πνεύμα συνεργασίας και με τις τροπολογίες σας ευελπιστώ ότι θα συγκεντρώσουμε πολιτική συνένεση και θα γίνουμε κέριος ε, διαπραγματευτικός και θα έχουμε ισχύσει διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο. Σε ό,τι αφορά το CF, τη διευκόλυνση του Connecting Europe, συνδέοντα την Ευρώπη. Ναι, μεν να μεταφερθούν κονδύλια από το Ταμείο συνοχή. αλλά όπω είπα και το πρωί και για τον κύριο Πακέ τη Γενική Διεύθυνση MOVE, αυτό θα το δεχόμαστε μόνο υπό όρου αυτή τη μεταφορά. Θα πρέπει ε, να είναι έτοιμα τα κράτη-μέλη, γιατί θα γίνει ε, θα υπάρξει μεγάλη αντιπαράθεση στο Συμβούλιο, θα πρέπει να κλιμακωθεί αυτή η διαμάχη. Καλό θα ήταν λοιπόν να συμπληρωθούμε για να ελοπίσουμε αυτό το στόχο και όταν συντρέξουν όλες οι προϋποθέσεις τότε θα μπορέσω και εγώ να καταθέσω συμβαστικές τροπολογίες και να συνεργαστούμε για να καταθέσουμε τέτοιες συμβαστικές τροπολογίες ώστε να είμαστε έτοιμοι για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού. Ευχαριστώ για την υπομονή σας. Κυρία Περνάμε τώρα στους κοιόδης εισηγητές το ΕΛΚ, κύριε Ματσόνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ με τον συνάδελφο Μποστινάρο και είμαι διατεθειμένη να γκρίνω, να δεχτώ μάλλον την πρόταση την οποία παρουσιάζει η Επιτροπή αν και θα πρέπει να ανοιχτούμε λίγο προς μια μελλοντική τροπολογητική δραστηριότητα θα έλεγα η οποία θα μας επιτρέψει να συμπεριλάβουμε θέματα τα οποία σε αυτή την πρώτη πρόταση δεν περιλαμβάνονται τουλάχιστον όπως τα θέλαμε και αναφέρομαι σε θέματα των μεταφορών στο Ταμείο για τις Μεταφορές το θέμα της αναφοράς της συμπερίληψης μάλλον της Natura 2000 κάτι το οποίο με τον τρόπο με τον οποίο είχε πεταθεί δεν ήταν ο σωστότερος και ειδική αναφορά στις ε, περιοχές της τα κτλ. Γενικά όλα αυτά όμως ε, μπορεί σε αυτή τη φάση που είναι μια φάση δεκτική, μια φάση ανοίγματο μπορούν να τεθούν στο μέλλον και να οδηγηθούμε σε σωστά αποτελέσματα. Θα ήθελα να κάνω τώρα λίγα σχόλια για την συζήτηση που έγινα σήμερα το πρωί και στην οποία δυστυχώς δεν μπόρεσα να πάρω μέρος. Θα ήθελα να συμφωνήσω με τους συναδέλφους που εξετίμησαν θετικά τις ε, εργασίες των την εργασία των Βανίς ρόι και της Κρέλα και τις οποίες είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε και στο παρελθόν δεν συμφωνώ με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που άκουσα και το απόγευμα για τη μακροοικονομική αιρεσιμότητα. Νομίζω ότι στο θέμα αυτό ίσως θα μπορούσαμε να επιστρέψουμε στις συγκεκριμένες προβλέψεις του Ταμείου Συνοχής και να δούμε ακριβώς τι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια γύρω από τον τρόπο λειτουργίας του. Έχει πάντως μεγάλη σημασία αυτό το οποίο λέγουν οι δύο εισηγητές για το γενικό κανονισμό. Διευκρινίζουν ότι θα πρέπει να ορίσουμε καλύτερα τις συμβάσεις εταιρικής φύσης, θα πρέπει να είναι ενισχυμένου τύπου και διευκρινίζουν επίσης ότι θα πρέπει επιτέλους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσπαθήσει να βρει τους τρόπους με τους οποίους να φύγουν κάποιοι κατάλογοι σε σχέση με τα ονόματα των πόλεων και να μιλήσουμε γενικότερα για μια πλατφόρμα στρατηγική που να καλύπτει το σύνολο των αστικών περιοχών και όχι μια λίστα με επιμέρους ονόματα που μπορεί να μην είναι πλήρης. Και εδώ υπάρχει ίσως χώρος και για την πρόταση του κυρίου Μποστινάρου είναι κάτι το οποίο άπτεται σαφώς των δημογραφικών πλευρών του θέματος που τέθηκε από τους εισηγητές και που θα πρέπει να υπογραμμιστεί ακόμα περισσότερο σχετικά με τις πολιτικές ανάπτυξης και τις πολιτικές συνοχής τις οποίες θέλουμε εμείς να πετύχουμε. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να παρατηρήσω εδώ ότι ο εισηγητής κατάφερε να εντοπίσει σωστά τις πιο σημαντικές πλευρές της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να βρει την ουσία με λίγα λόγια. Μας κάνει ο κ. Μποστινάρο ορισμένε προτάσεις με τις οποίες συμφωνώ. Θα πρέπει επίσης να συμπληρώσουμε όμως με κάποιο τρόπο τις προτάσεις του κυρίου Μποστινάρου. Νομίζω σχετικά με τις προτάσεις της Επιτροπής ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε κατά κάποιο τρόπο να διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογής του Ταμείου Συνοχής έτσι ώστε να μπορεί το Ταμείο Συνοχής να υποστηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως επίσης και τις επενδύσεις στον τομέα της κατάρτισης και της επιμόρφωσης. Αυτό είναι κάτι το οποίο ανταποκρίνεται στη στρατηγική 2020 και αυτό είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει στην σωστότερη χρήση της διαχείρισης του Ταμείου Συνοχής. Υποστηρίζω λοιπόν την πρόταση η οποία γίνεται για τη συμπερίληψη των δικτών ποιότητας οι οποίοι να στρέφονται, να προσανατολίζονται προς τα αποτελέσματα να συμπεριλάβουμε δείκτες οι οποίοι φυσικά να καλύπτουν τα θέματα της αηφορίας στην ανάπτυξη όπως ακριβώς είπε και ο κύριος Μποστινάρο και όπως το δείχνει και πιο συγκεκριμένα με τις τροπολογίες του. Όπως και για το ΦΕΝΤΕΡ τότε θα πρέπει και στο Ταμείο Σύνοχης να υπάρξει δυνατότητα βελτίωσης των υποδομών για να διευκολύνουμε έτσι την πρόσβαση στις βασικές υπηρεσίες και αναφέρομαι σε κάποιες συλλογικές μορφές υπηρεσίες όπως σαν παράδειγμα η κοινή θέρμανση των κατοικιών που είναι κάτι το οποίο χαρακτηρίζει ίσως περισσότερο κάποιες χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης και να προσπαθήσουμε να δούμε ε, σε αυτές ιδιαίτερα τις χώρες ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες. Τα προγράμματά μας λοιπόν θα πρέπει να έχουν ε, επίσης σαν στόχο την προώθηση της πράσινης ενέργειας και την βελτίωση της ενεργειακής αποτελεσματικότητας. Σχετικά τώρα με τον κατάλογο των προτεραιοτήτων και με τις κατά προτεραιότητα επενδύσεις. Εδώ θα πρέπει να προσθέσουμε σε αυτό τον κατάλογο των προτεραιοτήτων τουλάχιστον μία ακόμη η οποία μου φαίνεται ότι είναι πολύ σημαντική. Είναι η προώθηση των νέων τεχνολογιών, των αναδιωμένων τεχνολογιών που μπορούν να βοηθήσουν στην δημιουργία μιας οικονομίας με χαμηλές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω ότι στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γίνεται μία αναφορά στο ότι ε, τα προγράμματα τα οποία ε, χρηματοδοτούνται πιθανώς από το σύστημα ανταλλαγής ποσοστώσεων είναι κάτι ενός στις εκπομπές καυσαερίων είναι κάτι το οποίο δημιουργεί σύγχυση. Θα πρέπει το σύστημα αυτό με κάποιο τρόπο να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα και θα πρέπει τα σχέδια αυτά τα οποία χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα ανταλλαγής ποσοστώσεων ε, να είναι επιλέξιμα. Ο κύριος Χρυσόγελος. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τον εισηγητή, τον κύριο Μποστινάρου, γιατί είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία. Ε, στην έκθεσή του εντοπίζονται πραγματικά ε, τρία σημεία στα οποία συμφωνώ και μισό στο οποίο απλώς θα το επεκτείνω και σε κάποια άλλα που θα θέλαμε να έχουμε ορισμένες περισσότερες συζητήσει και προσθήκες. Είναι πολύ σημαντικό, νομίζω, και το αποδεχόμαστε να υποστηριχθεί η ένταξη των κατοικιών στο πεδίο εφαρμογή του κανονισμού για το Ταμείο Συνοχή, για να προωθεί η ενεργειακή απόδοση και ανανόσιμε πηγέ ενέργεια και στον τομέα αυτό. Είναι μια πραγματικά οικονομικά αποδοτική δυνατότητα να μειωθούν οι εκπομπέ ε, των αερίων θερμοκηπίου στι χώρε συνοχή και αυτό μπορεί να γίνει σε συνδυασμό με την δημιουργία θέσεων εργασία και την καταπολέμηση τη ενεργειακή φτώχεια. Δηλαδή, άνθρωποι που δεν έχουν να πληρώσουν λογαριασμού ε, θέρμανσης, ψήξης και ηλεκτρισμού. Επίσης είναι πολύ σημαντικό πιστεύω ε, για τη γενικότερη αηφορία και την επίτευξη της συνοχής η ένταξη των περιοχών Natura 2000 επενδυτικές προτεραιότητες του Ταμείου. Ευχαριστούμε τον κύριο Παστινάρου που το <laughs> συμπεριέλαβε. Είναι σημαντικό, σημαντικές αυτές οι περιοχές για την ποιοποικιλότητα μια και αντιπροσωπεύουν και το 20% τελικά της, ε, του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στα θέματα αυτά. Ε, η χρηματοδότηση αφορά την προστασία, διαχείριση και αποκατάσταση. Και αποκατάσταση έτσι κι αλλιώ η χρηματοδότηση σε αυτού του τομεί είναι περιορισμένη. Επίση, θεωρούμε πολύ σημαντικό ότι ε, λαμβάνονται υπόψη τα δικαιώματα των ανθρώπων που έχουν κινητικά προβλήματα. Αυτό πρέπει να περάσει σε όλου του κανονισμού και γενικά σε όλε τι πολιτικέ που περνάνε από το Κοινοβούλιο. Ε, και το τέταρτο, στο οποίο συμφωνούμε απόλυτα, είναι να περιληφθεί και το θέμα της υπαίθρου, δηλαδή το θέμα του περιβάλλοντος της υπαίθρου. Θα έλεγα, επειδή έχω και ένα ιδιαίτερο <laughs> ενδιαφέρον, επειδή κατάγμα από νησιά, ε, χωρίς να αποκλείεται και το θέμα των νησιών. Δηλαδή η βελτίωση και του νησιωτικού, του νησιωτικού περιβάλλοντος και των πόλεων που είναι σε νησιά, αλλά και γενικότερα του γύρω περιβάλλοντος. Θα θέλαμε να ε, δώσουμε λίγο μεγαλύτερη έμφαση σε ορισμένου τομεί, όπω για παράδειγμα το θέμα τη. ε, ενίσχυση ικανότητα των δημόσιων φορέων. Σε αυτό πρέπει να περιλαμβάνεται, το λέγαμε και το πρωί, και οι περιφερειακή φορείς και οι τοπικοί φορείς και η τοπική αυτοδιοίκηση και οι τοπικοί φορείς. Είναι πολύ σημαντικό γιατί ε, αν δεν ενδυναμώσει η ικανότητά τους τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην παρακολούθηση, εφαρμογή και αξιολόγηση δράσεων που γίνονται στις περιοχές τους, δυστυχώς δεν θα έχουμε αποτέλεσμα. Και σε αυτό νομίζω θα πρέπει να δώσουμε πολύ μεγαλύτερη έμφαση υπάρχουν αναφορές, αλλά πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση. Ε, το δεύτερο που θα πρέπει να δώσουμε λίγο μεγαλύτερη έμφαση, το λέγαμε και το πρωί, είναι να βρούμε την κατάλληλη ορολογία έτσι ώστε πράγματι ε, στα, στις εταιρικές συμβάσεις οι περιφέρειες να συμμετέχουν στην διαμόρφωση των σχεδίων. Δηλαδή είναι σημαντικό να βρούμε την κατάλληλη διατύπωση έτσι ώστε να μην παραμένει ω μια ευχή, γιατί ξέρουμε και από το παρελθόν τι έχει γίνει και ξέρουμε ότι μερικέ χώρε δεν έχουν παράδοση, θα λένε ναι, θα κάνουμε τη διαβούλευση, αλλά στην πραγματικότητα θα επεξεργάζονται μόνε του τα σχέδια που αφορούν περιοχέ. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε τρόπο, είτε μέσα από τον κώδικα συμπεριφορά, είτε μέσα από την ε, σαφή διατύπωση για συναπόφαση με το κράτος μέλος, τουλάχιστον για εκείνες τις δραστηριότητες, για εκείνα τα σχέδια που αφορούν συγκεκριμένες περιοχές. Δηλαδή περιοχές, περιφέρειες, αυτές που θα επηρεαστούν από τα σχέδια πρέπει να έχουν συναποφασίσει, να έχουν ε, με δεσμευτικό τρόπο συμμετάσχει στη διαδικασία. Στο θέμα των μεταφορών ε, θα θέλαμε να ε, πούμε ότι πρέπει να δοθεί έμφαση σε υποδομές μεταφορών που ε, ενισχύουν το συνδυασμό βιώσιμων συστημάτων μεταφοράς ε, και βιώσιμης κινητικότητας γενικότερα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και μέσα στις πόλεις αλλά και άλλες υποδομές που δεν είναι μόνο αυτοκινητόδρομοι, δεν είναι μόνο τρένο, είναι περπάτημα, ποδήλατο, μέσα μαζικής μεταφοράς, car sharing, pooling κλπ. Άρα να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση σε αυτό που είναι πιο βιώσιμο σε επίπεδο Τώρα, στο θέμα των δικτών, πράγματι έγινε και συζήτηση, αναφέρει και ο εισηγητή. Πρέπει να βρούμε πιο κατάλληλου δείκτε, γιατί αν η απόδοση αφορά πόσα χιλιόμετρα έγιναν ή πόσα χρήματα απορροφήθηκαν, αυτό δεν μπορεί να περιγράψει πραγματικά σήμερα πλέον τη συνοχή ή την περιφερειακή ανάπτυξη. Πρέπει να βρούμε κατάλληλου δείκτε που να ανταποκρίνονται σε αυτό που στάμε και εδώ, στην απόδοση, απόδοση σε θέματα συνοχή, σε θέματα εφορία και όχι μόνο απλώ δείκτε ποσοτικού που νομίζω δεν μα ε, αντιπροσωπεύουν πια. Στα θέματα τη προώθηση πυρηνική ενέργεια θα πρέπει να εξαιρεθεί πλήρω από το πεδίο εφαρμογή του Ταμείου Συνοχή και νομίζω θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη έμφαση έτσι ώστε τα έργα να μην κατευθύνονται ακόμα προ του ε, οδικού άξονε, σε οδικέ υποδομέ, ε, εξαίρεση ίσω αν υπάρχουν διασυνοριακέ συνδέσει, αλλά κυρίω σε τρένα και σε τέτοιε κατευθύνσει. Τώρα, στο θέμα των εγκαταστάσεων ε, τηλεθέρμανσης και τηλεψήξης είναι κάτι που νομίζουμε ότι θέλει περισσότερη συζήτηση. Υπάρχει, υπάρχουν δύο προβλήματα. Το ένα είναι ότι αυτές οι εγκαταστάσεις έχουν συμπεριληφθεί στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών και υπάρχει περίπτωση, εάν περιληφθούν σε αυτές τις χρηματοδοτήσεις, να ε, δημιουργήσουν προβλήματα στην αγορά ETS. Και το δεύτερο είναι ότι μην δοθεί λάθος μήνυμα για το θέμα των ανανώσιμων πηγών ενέργειας Εκεί νομίζω θα πρέπει να το συζητήσουμε ακόμα περισσότερο ε, και κλείνω λέγοντας αυτό που είπα και το πρωί. Ε, υπάρχει ένα θέμα ποια στατιστικά στοιχεία θα χρησιμοποιήσουμε για να κρίνουμε αν ένα κράτος, αν ένα κράτος μέλος είναι επιλέξιμο για το Ταμείο Συνοχής. Ε, η οικονομική κρίση και τα μέτρα λιτότητας έχουν αλλάξει πάρα πολλά δεδομένα. Πρέπει να είναι όσο πιο πολύ μέσα η περίοδος της κρίσης. Και αυτό θα πρέπει να το διευκρινίσουμε ε, έτσι ώστε πραγματικά να λάβουμε υπόψη ότι η κρίση έχει αλλάξει πάρα πολλά πράγματα χωρίς να παραγνωρίζουμε τα κράτη που ήταν έτσι και αλλιώ, βέβαια σε δυσμενέστερη κατάσταση και πριν την κρίση. Ευχαριστώ πολύ. Η Κορνίδια <clears throat> δεν είναι παρούσα. Και εγώ, λέει ο έχω λάβει μια, ένα ταχυδρομείο που μου τονίζει την ε, ε, υποστήριξη του σχεδίου, ε, κυρία Έρνστ. Και τώρα προχωρούμε στους άλλους αγορητές, Τόμας Πρέμπα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα εν συντομία να πω ότι Συμφωνώ με την προσέγγιση του εισηγητού για το Ταμείο Συνοχής. Η ομάδα μου, οι μεταρρυθμιστές ε, και συντηρητικοί, ενστερνίζονται γενικώ στις προτάσεις του εισηγητού. Υπάρχουν βέβαια κάποια θέματα που μας ενοχλούν και γι' αυτά θα καταθέσουμε τροπολογίες. Ε, ξέρουμε ότι εσείς είστε υπέρμαχος ε, της ε, διευκόλυνση του μέσου του Connecting Europe. Εμείς αντίθετα είμαστε κατά αυτού του μέσου. Ούτε είμαστε υπέρ της μεταφοράς ε, του το κονδυλίων από το Ταμείο Συνοχής στο Connecting Europe. Αν γίνει μεταφορά γίνει πολύ μικρότερη και προτιμούμε και καθόλου. Γιατί το Connecting Europe ουσιαστικά μειώνει τη, τα εθνικά μερίδια από το Ταμείο Συνοχής και προσωπικά πιστεύω αλλά και η ομάδα μου πιστεύω ότι καλύτερα θα μπορούσαν τα κονδύλια αυτά να τα εκμεταλλευτούν στο πλαίσιο του Ταμείου Συνοχή στα κρατημέλη και όχι με το Connecting Europe, με το Συνδέοντα την Ευρώπη. Μα προβληματίζει κάπω και η μεταφορά κονδυλίων από την πολιτική συνοχή στα θεματικά ταμεία, το Ταμείο Μεταφορών, και άλλα γιατί γίνεται κεντρική διαχείριση από τις Βρυξέλλες και δεν μας ε, βρίσκει και πολύ σύμφωνος κάτι τέτοιο. Για πολλά θέματα ε, η πολιτική συνοχής ε, δεν εξυπηρετείται από κεντρική διαχείριση των θεματικών αξώνων από τις Βρυξέλλες. Επίσης, σε ό,τι αφορά τη μετάβαση σε μια οικονομία με χαμηλή χρήση άνθρακα. Προτιμώ να μιλούμε για οικονομία με χαμηλές εκπομπές αερίου του θερμοκηπίου και όχι χαμηλή χρήση άνθρακα. Έχουμε πολλά επιχειρήματα υπέρ αυτής της προσέγγισης, γιατί πρώτα θα έχει τεράστιο κόστος η μετάβαση σε μια οικονομία με χαμηλή χρήση άνθρακα. Για αυτά τα τρία σημεία που σας ανέφερα θα καταθέσουμε συγκεκριμένες τροπολογίες και θα προσπαθήσουμε να μεταπίσουμε τον εισηγητή, ώστε τουλάχιστον ένα τμήμα των παρατηρήσεών μας να, τα, να τις λάβει υπόψη. Ευχαριστώ, ο Σον Κέλλη. Firstly, thanks to the rapporteur as well. I think he gave a very practical summary of... Uh, Βλέπουμε λοιπόν σε ποια φάση βρισκόμαστε με πρακτικό τρόπο Υπάρχουν δύο τομείς βέβαια στους οποίους ε, έχουμε πολλά να κάνουμε ιδιαίτερα στα πλαίσια της εποχής αυτής λιτότητας και ύφεση. Ο ένας τομέας είναι η εκπαίδευση, δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε αυτό. Αν θέλουμε πράγματι να προχωρήσουμε οικονομικά, η εκπαίδευση και η κατάρτιση είναι απαραίτητες. Και δεύτερον η ενέργεια, Έχουμε τους στόχους του 2020, έχουμε στόχους επίσης και στο, για το 2050 στον τομέα και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να υπογραμμίσουμε τη σημασία των επενδύσεων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών. Και νομίζω ότι άλλοι έχουν πετύχει πολύ περισσότερα από εμά και θα πρέπει να τους μιμηθούμε. Γι' αυτό λοιπόν ακούσαμε ευχαρίστηση της προτάσεις του εισηγητή. Θυμίζω επίσης ότι εδώ στο Κοινοβούλιο είχαμε και μία παρουσίαση υψηλού επίπεδου για το φυσικό αέριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για τις πιθανές προκλήσεις και δυσκολίες που μπορεί να έχουμε. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολεί. Όσο περισσότερο μπορούμε να παράγουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο το καλύτερο για την οικονομία. Και δεύτερον, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και με το υγροποιημένο φυσικό αέριο, τι γίνεται με το μεθάνιο προπάνιο και με κάποιες ε, επίσης ε, δραστηριότητες ε, για την σύλληψη των αερίων, την εξαγωγή και σύλληψη των αερίων, κάτι το οποίο μπορεί να δημιουργήσει ίσως κάποια προβλήματα και είναι κάτι το οποίο δημιουργεί διαφωνίες. Πάντως έχουμε πολλά να πετύχουμε με το αέριο ε, μη βλάπτοντας το περιβάλλον ή βλάπτοντας σε πάση περιπτώσει λιγότερο το περιβάλλον. Και νομίζω ότι εδώ αν μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις υποδομές γύρω από το αέριο θα διευκολύνουμε τους στόχους μας για το 2020, θα αναπτύξουμε μια οικονομία ιδιαίτερα φιλόδοξη ε, και θα γίνουμε ουσιαστικοί και σημαντικοί στον κόσμο όχι μόνο λοιπόν για την Ευρώπη δεν είναι σημαντική αυτή η δραστηριότητα αλλά και για τη θέση μας στον κόσμο. Ο κύριος Σόλμπριχτ. Θα ήθελα να υπογραμμίσω κάποια από τα σημεία τα οποία τέθηκαν ήδη. Πρώτον, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το ξεκάθαρο μήνυμα το οποίο αποστέλει. Νομίζω ότι είδαμε κατά τη διάρκεια της συζήτησης ότι υπάρχουν αρκετές παρανοήσεις γύρω από τα θέματα αυτά. σε σχέση με το συγκεκριμένο τομέα είναι κατά του Connecting Europe. Ίσως εδώ να υπάρχει κάτι το οποίο χρήζει περισσότερο διευκρίνησης μεταξύ μας, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι μια εξαίρεση. Αυτό το οποίο συζητάμε τώρα είναι το Ταμείο το οποίο αφορά ουσιαστικά ένα τμήμα της Ευρώπης και αυτό πρέπει να μην το ξεχνάμε. Είναι για τις χώρες συνοχής το Ταμείο αυτό και υπολογίζεται το ποσοστό του ανώτερο σε ΝΑΤΣ2, δηλαδή σε εθνικό ουσιαστικά επίπεδο, και δεύτερον αντιμετωπίζεται όχι σαν ένα περιφερειακό ταμείο, αλλά σαν ένα εθνικό ταμείο. Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό του. Εξορισμού λοιπόν είναι κάτι το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε, ευρωπαϊκό, περιφερειακό συγγνώμη, επίπεδο αλλά έχει σχεδιαστεί επί τη βάση δεδομένων που έχουν συλλεγεί σε εθνικό επίπεδο. Αυτή είναι η πραγματική διαφορά ανάμεσα σε αυτό το ταμείο και τα διαφθορτικά ταμεία. Το να ενισχύσει τις περιφέρειες κανείς μέσω αυτού του ταμείου είναι κάτι το ενδιαφέρον, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί γιατί όπως είπα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο και μιλάμε και για χώρες οι οποίες δεν έχουν περιφέρειες με την έννοια που εμείς δίνουμε στις περιφέρειες. Η Ουγγαρία σαν παράδειγμα. Δεν έχουν διοικητικές δομές που να ονομάζονται περιφέρειες. Ενώ η Ρουμανία έχει σαν παράδειγμα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα σημείο, είναι τα ειδικά χαρακτηριστικά του Ταμείου. Αυτό που έχει επίσης σημασία είναι ο τρόπος με τον οποίο συνδέεται το συγκεκριμένο Ταμείο και οι υποδομές και το πρόβλημα των υποδομών στις πιο αναπτυγμένες χώρες. Και ίσως εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορεί λίγο να μας διαφωτίσει. Στη δική μου έκθεση η οποία ασχολείται πολύ στενά με τα θέματα της συνοχής, υπάρχει ένα άρθρο το οποίο λέει ότι για τις βασικές υπηρεσίες, για τις επενδύσεις στις βασικές υποδομές, στις μεταφορές, στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες κτλ. Το τονίζουμε αυτό. Γιατί? Γιατί ακριβώς υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης. Κάτι δηλαδή το οποίο μπορεί να επενδυθεί από το Ταμείο αυτό στις χώρες συνοχής είναι κάτι το οποίο μπορεί και να μην μπορεί να γίνει στις πιο αναπτυγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά αυτό αντίστοιχα που δεν είναι επιτρεπτό μπορεί να γίνει επιτρεπτό μέσω του Connecting Europe. Πρέπει να είμαστε λοιπόν προσεκτικοί σε σχέση με το τι ζητούν οι χώρες αυτές. Οι επενδύσεις αυτές οι οποίες θα προέλθουν από το Ταμείο Συνοχής και θα μεταφερθούν ουσιαστικά προς το Connecting Europe δεν ξέρουμε αν είναι κάτι το οποίο μπορεί να λειτουργήσει στις ε, αναπτυγμένες περιφέρειες ή τις αναπτυγμένες χώρες. Λοιπόν, τι έχουμε να κάνουμε εδώ τώρα. Έχουμε ένα κομμάτι εδώ του Connected Europe χωρίς ε, το Ταμείο Συνοχής. Αυτό ισχύει για λίγες χώρες, για συγκεκριμένες χώρες ή έχουμε να κάνουμε κυρίως για υποδομές ε, στον τομέα της ενέργειας και των μεταφορών. Δεν είναι διόλου τυχαίο που ο εισηγητής συνέδεσε το Ταμείο Συνοχής και την ενέργεια. Είναι ασυνήθες αυτό το οποίο έκανε. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι εύκολο για να διευκρινιστεί. Εμείς είχαμε συμπεριλάβει το θέμα σαν παράδειγμα της ενεργειακής αποτελεσματικότητας στα κτίρια. Αν το συμπεριλάβουμε και στο Ταμείο Συνοχής, τότε θα πρέπει να διευκρινίσουμε με διαφορετικό τρόπο το τι είδους χρήματα θα πάνε στο ένα ταμείο και τι χρήματα θα πάνε στο άλλο ταμείο. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο όταν συζητούσαμε για το Connecting Europe θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο να παίρνουμε χρήματα από τους εθνικούς φακέλους και να τα βάζουμε σε ευρωπαϊκές υπηρεσίες. Αλλά τι γίνεται με το σύνδεσμο ανάμεσα στα υπόλοιπα του Connecting Europe, την ενέργεια, την ενημέρωση και με την απαγόρευση ουσιαστικά ε, η οποία υπάρχει για χρήματα που προέρχονται από το Ταμείο Συνοχής να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των υποδομών στις προχωρημένες χώρες ή στις πιο αναπτυγμένες χώρες. Λοιπόν, ε, είδαμε με το παράδειγμα ε, της Ουγγαρίας Είδαμε επίσης και το τι λέει η συνθήκη του Μάστριχτ, η οποία συνιστά στη συγκεκριμένη περίπτωση μια μακροπεριφερειακή κύρωση σήμερα. Είναι κάτι το οποίο μόλις έχει αρχίσει να ισχύει στην Ουγγαρία. Πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί τώρα να διευκρινίσουμε αυτά τα πράγματα να ξεκαθαρίσουμε ότι είμαστε κατά της, α, ε, α, ε, της ε, μακροπεριφερειακής αιρεσιμότητας λέει ο μιλητής ενώ στην συνοχή υπάρχει, μια, υπάρχει ίσως μια πιθανότητα σύγχυσης σε πάση περιπτώσει με το Περιφερειακό Ταμείο δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά εδώ υπάρχει το θέμα της σχέσης με τις πιο αναπτυγμένες χώρες, ακόμα όπως είπα και αν και το Ταμείο Συνοχής δεν προορίζεται για αυτούς. Έχει το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Director General, the floor is yours. <laughs> Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το πολύ αξιόλογο έργο του, τη γνωμοδότησή του επί της προτάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Ταμείο Συνοχής. Χαίρομαι που υποστηρίζει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς τα βασικά στοιχεία της τουλάχιστον. Δύο είναι τα κυρία θέματα που προκύπτουν από τις τροπολογίες και που συζητήσαμε το απόγευμα. Το πρώτο αφορά το τι μπορεί να καλύπτει το Ταμείο Συνοχής και τι εκπίπτει το Ταμείο Συνοχής και την τροπολογία που προβλέπει επέκταση ώστε να καλυφθεί η συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας ψήξης, η θέρμανση και ψήξη της πόλης κτλ. Επίση μία συνέπεια σε ό,τι αφορά τη χρήση των κοινοτικών κονδυλίων. Υπάρχουν ε, δυνατότητε διευκρίνηση διευκρίνησης ε, στην πρόταση του τι θα χρηματοδοτείτε και τι όχι. Πάντως, η Επιτροπή φρονεί ότι τα κοινοτικά κονδύλια και η χρήση του Ταμείου Συνοχής δεν θα πρέπει να υπονομεύουν <clears throat> την αποτελεσματικότητα του συστήματος εμπορίας εκπομπών. Οπότε μία τροποποίηση που επιτρέπει στο Ταμείο Συνοχής να στηρίξει επενδύσεις σε εργοστάσεις, σε εγκαταστάσεις που καλύπτονται από το σύστημα εμπορίας εκπομπών είναι κάτι παράλογο κατά τη γνώμη μας γιατί υπονομεύει ένα μηχανισμό το σύστημα εμπορίας εκπομπών που στόχο έχει τη μείωση των καυσαέριων. Ως εκ τούτου δεν έχει νόημα για μας. Βέβαια δεν αποκλείεται όπως είπα, να γίνουν κάποιες διευκρινήσεις της διατύπωσης, ώστε να αποσαφινιστεί ότι οι συναφείς υποδομές μπορούν να τύχουν χρηματοδότησης. Τώρα, σε ό,τι αφορά πάλι το τι χρηματοδοτεί και τι όχι το Ταμείο Συνοχής, ε, αφορά την επέκταση των επενδύσεων που αφορούν την ενεργειακή αποδοτικότητα και στον τομέα της στέγασης. Συμφωνούμε με τη σημασία που έχουν οι επενδύσεις στην ενεργειακή αποδοτικότητα, κύριε Μποστινάρου, αλλά θεωρούμε ότι καλό θα ήταν να διαχωρίσουμε τον προορισμό των διαφόρων ταμείων, των κονδυλίων των διαφόρων ταμείων. Έγιναν κάποιες αλλαγές μεταξύ της διάκρισης ε, ΦΕΝΤΕΡ και Ταμείου Συνοχής, και, αλλά πιστεύω ότι ο προορισμός του Ταμείου Συνοχής είναι σαφής και κατοχυρώνει και τη συνθήκη. Στηρίζει τα διευρωπαϊκά δίκτυα και περιβαλλοντικά προγράμματα, ε, κυρίως ε, με έμφαση το περιβαλλοντικό κεκτημένο. Βέβαια, δεχόμαστε κάποια ελαστικότητα στην εφαρμογή, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να κρατήσουμε μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ των ταμείων και πιστεύω ότι είναι σωστή διαχωριστική γραμμή της πρότασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, δεν δικαιολογείται και από τις ανάγκες να ενισχύσουμε τη χρηματοδότηση των κρατών μελών ε, από τα κονδύλια του ΦΕΝΤΕΡ προκειμένου να καλύψουν τις επενδυτικές ανάγκες για την ενεργειακή αποδοτικότητα των σπιτιών. Γιατί έτσι μπορεί να αλλοιωθεί ή να υποβαθμιστεί η αποτελεσματικότητα του Ταμείου συνοχή και να μην χρησιμοποιούνται τα κονδύλια του Ταμείου συνοχή για το βασικό του προορισμό που κατοχυρώνεται, όπω είπα, και από τη συνθήκη. Γι' αυτό και έχουμε επιφυλάξεις ως προς τη συγκεκριμένη πρόταση του εισηγήτου. Τώρα μερικά άλλα θέματα. Σε ό,τι αφορά τη μνήα του Natura 2000, στην τροπολογία 8 δηλαδή, πιστεύουμε ότι είναι περιττή ε, η διατύπωση, προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας. Ούτως ή άλλως ε, η προσέγγιση μας είναι ευρύτερη. Ένας περιορισμός τους δημιουργεί σε ερμηνευτικά προβλήματα. Είναι περιττή αυτή η προσεγγιση μας ειναι ευρυτερη ενας περιορισμος τους δημιουργει κατά τη γνώμη μας. Σε ό,τι αφορά την προσθήκη της μίας της προσπελασιμότητας, της τροπολογίας 10 και 11, επί της αρχής συμφωνούμε με τον εισηγητή, αλλά όπως θα ξέρετε το θέμα αυτό καλύπτεται στις εξάντε ρεσιμότητες του παραρτήματος 4 του κανονισμού με τις ε, κοινέ διατάξει. Υπάρχει μια γενική προκαταρκτική αιρεσιματικότητα, η αιρεσιμότητα σχετικά ιδιαίτερα με την προσπελασιμότητα. Και αυτό σε σχέση με συγκρίσιμες επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από το ΦΕΝΤΕΡ. Πάντως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ταχθεί υπέρ τη διατήρησης αυτής τη προκαταρκτική αιρεσιμότητα για να υπάρχει διαβεβαίωση ότι όλες οι επενδύσει θα πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια της ε, πρόσβασης. Και τέλος, για το μέσο τη διευκόλυνση του συνδέοντας την Ευρώπη, το Connecting Europe Facility, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πρόθυμη και συνεργάσιμη θέλουμε συνέχεια του, συνέχιση του διαλόγου και με τον εισηγητή και με τους συναδέλφους της Γενικής Διεύθυνσης MOVE για να δούμε ποιοι μηχανισμοί είναι οι κατάλληλοι ώστε να εξασφαλίσουν τη χρήση των 10 δισεκατομμυρίων που μεταφέρονται στο μέσο Connecting Europe. Και πιστεύω ότι αυτό που μας ενδιαφέρει σήμερα είναι ο συνδυασμός του Ταμείου Συνοχής και του Connecting Europe αφορά τα 10 δισεκατομμύρια, τη μεταφορά των 10 δισεκατομμύριων. Στόχος είναι να χρησιμοποιηθούν για τις ίδιες επενδύσεις, για τις μεταφορές δηλαδή, όπως θα χρησιμοποιούνται και από το Ταμείο Συνοχής. Με στοχευμένο όμως τρόπο και με πλήρη, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις κοινοτικές ε, προ, προτεραιότητες. Ενώ το Connecting Europe στηρίζεται σε άλλες επενδύσεις, ε, προορίζεται για άλλες επενδύσεις. Και όπως είπε ο κύριος Όλμπριχτ, αυτό είναι ένα επιχείρημα που συνηγορεί υπέρ του περιορισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις βασικές υποδομές, στις, περισσότερα, στις πιο ανεπτυγμένες περιοχές. Βέβαια, υπάρχουν και άλλα επιχειρήματα κατά τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που συνηγορούν υπέρ του περιορισμού του της εμβέλειας της χρήση του ΦΕΝΤΕΡ για τις βασικές υποδομές σε πιο ανεπτυγμένες περιοχές. Και αυτό θα το συζητήσουμε αργότερα όταν θα εξετάσουμε τον κανονισμό για το ΦΕΝΤΕΡ, το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Αυτά προς το παρόν ως προς την ε, την έκθεση του κ. Μποστινάρου. Ευχαριστώ. Θέλετε να ολοκληρώσετε τη συζήτηση κύριε Μποστινάρο. Πρώτον, θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια θέματα τα οποία έθεσαν οι συνάδελφοι και μετά να αναφερθώ σε λίγα από τα σχόλια που έκανε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. από τον Γενικό Διευθυντή της ε, Διεύθυνσης Ρέντζιου. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Ματσόνη και νομίζω ότι η συνεργασία μας θα συνεχιστεί και θα συμπεριλάβει το τελικό αποτέλεσμα και άλλες σκέψεις οι οποίες είναι, σεβαστές, ε, είναι σύμβατες με τους στόχους του Ταμείου Συνοχής. Για την κυρία Μανέσκου, η ιδέα θα έλεγα για τη βοήθεια των μικρομεσαίων. Προφανώς οι προτάσεις μου είναι υπέρ των μικρομεσαίων ιδιαίτερα για την εξοικονόμηση ενέργειας στις κατοικίες, όπως επίσης και για τις εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας για θέρμανση και ψήξη. Οι κοινέ μονάδες παραγωγής ενέργειας θέρμανσης και ψήξης. Για τον κύριο Χρυσόγελο θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά για την εξαιρετική συνεργασία την οποία έχουμε μαζί τους Συμμερίζομαι αρκετέ από τις ανησυχίες σας, υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί όμως οι οποίοι διαφεύγουν των δυνατοτήτων και τη εμβέλειας του Ταμείου Συνοχής. Το Ταμείο Συνοχής δεν μπορεί να αντιμετωπίσει κάποια από τα προβλήματα στα οποία αναφερθήκατε. Πάντως λαμβάνουμε υπόψη αυτά που είπατε και συμφωνώ μαζί σα ότι και η διοικητική ικανότητα και η διοικητική ανάγκη η οποία υπάρχει για τις ε, συμβάσεις αυτές της εταιρική φύσης να βελτιωθούν ακόμα περισσότερο και να βελτιώσουν με τη σειρά τους την διοικητική δυνατότητα που έχουμε σε σχέση με αυτή τη μορφή παρέμβασης γιατί αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να βελτιώσει όχι μόνο τους ρυθμούς απορρόφησης αλλά και να βεβαιωθούμε ότι η μελλοντική μας πολιτική στον τομέα αυτό, η πολιτική συνοχή, θα ωφελήσει πράγματι τους πολίτες για τα σχόλια του επόμενου μιλητή Πορέμπας. Εγώ δεν είμαι φανατικός υπέρ του ΣΥΕΦ. E αντίθετα, κάποιοι θεωρούν ότι ε, σκέφτομαι ακριβώς αντίθετα από ό,τι σας λέω. Πάντως δεν είμαι ούτε άγγελος ούτε διάβολος. Η γνώμη μου, η οποία επιβεβαιώθηκε και από τον Νίκολας Μάρτιν, λέει ότι τελικά είμαι υπέρ του να δεχτώ τη δυνατότητα τα 10 εκατομμύρια τα οποία πρέπει να δοθούν μπορεί να υπάρξει αυτό. Είναι μια ανησυχία όπως είπε και ο κύριος Μάρτιν για τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη-μέλη θα μπορέσουν να δεχθούν την ιδέα να φύγουν τα δεκαδίς αυτά. Κάτι το οποίο θα μειώσει ουσιαστικά τα εθνικούς τους λογαριασμούς, φακέλους και δεν θα έχουν και τίποτα να πούν, δεν μπορούν να επηρεάσουν και τα έσοδα για την εφαρμογή των προγραμμάτων όταν εφαρμόζονται τα προγράμματα. Σχετικά με τα σχόλια τώρα του κυρίου Όλμπρεχτ και επιστρέφω πάντα στο Connecting Europe. Αυτό αναφέρεται στα διαμεθοριακά προγράμματα, έτσι δεν είναι. Ξέρετε πολύ καλά ότι αυτό το οποίο πιστεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι η συνεχισμότητα σε διαμεθοριακό επίπεδο δεν είναι αρκετά προχωρημένη και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να βελτιωθεί. Και γι' αυτό ακριβώς προτείνουμε να συνεισφέρει για την καλύτερη διασυνδεσιμότητα των κρατών μελών σε διαμεθοριακό επίπεδο και το Ταμείο Συνοχής. Η πραγματικότητα σε ορισμένες χώρες όμως ε, σαν την Πολωνία δείχνει το αντίθετο. Πάντως θα ήθελα να συνεργαστώ στενότερα και με τη Γενική Διεύθυνση MOVE έτσι ώστε να καλύψουμε τα κενά με τρόπο αποδεκτό από όλους και τα χρήματα τα οποία φεύγουν να επανέλθουν μέσω επενδύσεων σε αντίστοιχο περίπου όγκο, σε αντίστοιχη ποιότητα και ποσότητα και ταυτόχρονα τα κράτη-μέλη να έχουν κάτι να πούν, να έχουν λόγο εν περιπτώσει να αποφασίζουν και να εφαρμόζουν προγράμματα τα οποία να είναι θα έλεγα σύμβατα με τις απαιτήσεις ε, του Connecting Europe η βασική αρχή του όποιος κάνει πρώτος αίτηση αυτός παίρνει τα λεφτά θα πρέπει να απορριφθεί διότι δεν λαμβάνω υπόψη την ποιότητα εδώ και τον ανταγωνισμό. Έχει σημασία όμως να πούμε ότι το σύνθημα αν θέλετε της ε, πολιτικής συνοχής είναι η αλληλεγγύη. Καλός ο ανταγωνισμός αλλά πρέπει να συνδυάζεται από αλληλεγγύη. Κάποια κράτη-μέλη λοιπόν ανησυχούν γιατί, γιατί σήμερα δεν είναι σε θέση να προετοιμάσουν, να σχεδιάσουν και να προτείνουν στο pipeline της DG Move, της Γενικής Διεύθυνσης Move, κάποια προγράμματα τα οποία να είναι άμεσα επιλέξιμα. Και έχει ξεκινήσει μια συζήτηση ανάμεσα στην Γενική Διεύθυνση Move και στη Γενική Διεύθυνση Regio και ίσως κάποια στιγμή να επανέλθουμε στο θέμα μέσω μιας συμβιβαστικής τροπολογίας. Τώρα πάντα στα πλαίσια των σχολείων του κυρίου Μάρτιν. Η ιδέα αυτή δεν είναι αποκλειστικά δικείου. Για να συμπεριλάβουμε την ενέργεια δηλαδή για τις κατοικίες και την ενέργεια που απαιτείται για τα συλλογικά συστήματα θέρμανσης. Πολλές χώρες μέλη εκφράζουν την επιθυμία τους να χρησιμοποιήσουν και τα ταμεία συνοχής για τα συγκεκριμένους τομείς. Είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό για την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Είναι κάτι το πάρα πολύ... Other uh, type of And even more uh, Είναι κάτι το οποίο αφορά ορισμένες χώρες και για αυτές τις χώρες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει δυνατότητα ε, να χρησιμοποιηθούν ε, εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας τρίτης γενεάς οι οποίες ε, να μας επιτρέψουν να... Και αναφέρομαι πάντα σε θέματα ίσως που θα ονομάζαμε θέματα τηλεθέρμανσης ή συλλογικής κοινωνικής θέρμανσης. Πρέπει λοιπόν να υποστηρίξουμε τα κράτη-μέλη, να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν και το Ταμείο Συνοχής αν θεωρούν ότι αυτό είναι σημαντικό και είναι σημαντικό αν δει κανείς τι γίνεται σήμερα. Κοιτάξτε, σκεφτείτε τι συμβαίνει σήμερα. Σε πάρα πολλές χώρες μέλη θα πετύχουν τους στόχους του 2000, δεν θα πετύχουν μάλλον τους στόχους του 2020 και θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμα και ταυτόχρονα θα έχουν αποτύχει χωρίς να κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους, χωρίς να δώσουν κίνητρα για επενδύσεις σε χώρες όπως η Σλοβακία, η Ουγγαρία, η Πολωνία κτλ. Το θέμα είναι να βρούμε μια λύση σε σχέση με τα προβλήματα αυτά τηλεθέρμανσης και αν πράγματι θέλουν τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν και το Ταμείο Συνοχής για τη βελτίωση αυτών των συστημάτων να μπορούν να το κάνουν. Θα πρέπει εδώ να διευκρινίσουμε τα χρήματα που προέρχονται από το περιφερειακό και τα χρήματα που προέρχονται από το Ταμείο Συνοχής και δεν θα πρέπει να υπάρχουν επικαλύψεις. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να χρησιμοποιούν το Ταμείο Συνοχής και για την εξοικονόμηση ενέργειας στις κατοικίες. Κάτι το οποίο υπό τους υπάρχοντες κανόνες δεν είναι εφικτό και για το Natura 2000. Πράγματι θα πρέπει να χρημοσποιηθούν χρήματα για την αποκατάσταση και την προστασία της βιοπικιλότητας. Το Natura 2000 είναι ένας πολύ συγκεκριμένος χώρος, μάλλον πολύ πολύ συγκεκριμένοι χώροι, οι οποίοι μπορούν να γίνουν αντικείμενο διατήρησης με διαφορετικούς τρόπους. Και ξέρετε και ποια είναι η πραγματικότητα σήμερα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συστηματικά αποτυγχάνει τους στόχους τους οποίους έχει στο τομέα της, επικο... της ε, ε, Θα πρέπει να δείξουμε λίγο φαντασία εδώ και θα πρέπει να επιτρέψουμε έτσι ώστε ένα κομμάτι τουλάχιστον ε, που, με το, οποίο, το οποίο καλύπτει το Natura 2000 να βοηθήσουμε να λειτουργήσει σωστά. Έχω υπόψη μου τον, το, το δεκτικό του χαρακτήρα στο συγκεκριμένο κλάδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξέρω την αποφασιστικότητα και την ετοιμότητα της Προεδρίας, της Δανίας και υπάρχει και υποστήριξη από πλευράς του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και νομίζω ότι μπορούμε τελικά να πετύχουμε και να καταλήξουμε σε μια θετική πρόταση η οποία θα είναι ωφέλιμη για την πολιτική συνοχή και την εφαρμογή της στα επόμενα προγράμματα. Ευχαριστούμε κύριε Μποστινάρου. Ας περάσουμε στο σημείο 12 της, Ευρω... της διάταξής μας, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Η συγγήτριά μας είναι η κυρία Μαρία Ιρηγκογέν Πέρες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που εξετάζουμε τα ταμεία δίνοντας έμφαση και στους εργαζόμενους μέσω του Κοινωνικού Ταμείου και μέσω της γνωμοδότησής μου που ελπίζω ότι θα είναι έτοιμη στα αγγλικά τουλάχιστον το συντομότερο δυνατό προκειμένου να προβλέψουμε και διορία για την υποβολή τροπολογιών. Ε, που αν δεν κάνω λάθος ε, θα ξεκινήσει στις 8 Μαΐου. Θα κάνω μια σύντομη αναδρομή των ε, βασικών προσεγγίσεων της γνωμοδότησης και θα σας δώσω και κάποιες αδρές γραμμές των τροπολογιών. Προσβλέπω στη συνεργασία με τους συναδέλφους και στη βοήθεια των σκιωδών εισηγητών καθώς και στο διάλογο με τις ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις και τους εκπροσώπους κοινωνίας των πολιτών. Έτσι θα συμβάλλουμε στη δημιουργία μιας μεστής έκθεσης που θα καταλήξει στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της ελαστικότητας του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου θέλουμε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο να χρηματοδοτείται επαρκώς ώστε να υλοποιήσει τους στόχους του και να μετατραπεί σε ένα ουσιαστικό εργαλείο που θα βελτιώσει την ε, οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή περιορίζοντας τις ε, ανισότητες μεταξύ των περιφερειών και τις ανισότητες σε επίπεδα απασχόλησης μεταξύ τοπικού, περιφερειακού, και εθνικού επίπεδου. Επίσης μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία περισσότερων θέσεων απασχόληση, βελτιώνοντα την ποιότητα τη απασχόληση και ενισχύοντα ε, τα προσόντα και τα εφόδια των ε, εργαζομένων για να καλύπτουν τι ανάγκε και τι αγορά εργασία. Ό,τι αφορά ε, το πρόγραμμα επιστηστικής βοήθεια που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Θα ήθελα να ζητήσω από του εκπροσώπου Ευρωπαϊκή Επιτροπή περισσότερε πληροφορίε για το τι γίνεται και αν υπάρχει κάποια εξέλιξη ότι αφορά αυτή την πιθανότητα. Τέλο, ό,τι αφορά την ελαστικότητα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, θα ήθελα να τονίσω την ανάγκη η θεματική συγκέντρωση να είναι ελαστική για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα κονδύλια ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του κάθε κράτους μέλους και της κάθε περιφέρειας. Εγώ προτείνω ενίσχυση της ελαστικότητας του Κοινωνικού Ταμείου αυξάνοντας τις προτεραιότητες από 4 σε 6 σε περιφερειακό επίπεδο και μειώνοντας τα ποσοστά συγκέντρωσης. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των εταίρων, η συμμετοχή και των τοπικών και περιφερειακών αρχών, αλλά και των κοινωνικών φορέων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων, και σε τη φάση της ε, εκπόνησης, αλλά και σε φάση της εφαρμογής των μέτρων του Κοινωνικού Ταμείου και μάλιστα με συστηματικό και συγκροτημένο τρόπο και την δυνατότητα χρηματοδότησης αυτής της συμμετοχή, όχι μόνο με συνολικές επιχορηγήσεις, αλλά και με τη μορφή τεχνογνωσία είναι απαραίτητη. Έτσι, κάτι τέτοιο προβλέπεται στα άρθρα 108 και 109 του κανονισμού για τις κοινέ διατάξεις. Επιπλέον, θεωρώ ότι η πρόσβαση στα επιχορηγούμενα μέτρα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βελτιωθεί να βελτιωθεί η ικανότητα των κοινωνικών φορέων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων, δεν θα πρέπει να περιορίζεται στι μειονεκτικέ ή στι λιγότερο ανεπτυγμένε περιοχέ, ε, αφήνοντα ε, εκτό νυμφώνω στι μεταβατικέ περιοχέ που επίση ε, έχουν συμφέρον να προχωρήσει στον τομέα αυτό. Επίση θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε και μικρότερες περιφερειακές αρχές, ιδιαίτερα στις, στην Ήπεθρο, που δεν έχουν αρκετά μέσα και ικανότητα. Επίσης, θέλουμε μια ποσόστοση για την βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων. Θα πρέπει μέσω του Κοινωνικού Ταμείου να στηρίξουμε μια βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων με στρατηγική και ολοκληρωμένες δράσεις, ώστε να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αστικές περιοχές που περιλαμβάνονται στη Σύμβαση Σύνδεσης. Θα καταθέσω και τροπολογίες προκειμένου να συμπληρώσω κάποια, κάποιες πτυχές όπως τη συμπερίληψη της ισότητας ευκαιριών, ε, την αποφυγή των διακρίσεων, την προσαρμογή των μέτρων στις ιδιαίτερες ανάγκες των πιο μειονεκτικών ομάδων και την ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι μειονεκτικές περιοχές και κοινότητες. Επίσης, ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι σκοπός μου είναι τουλάχιστον στα αγγλικά να είναι έτοιμη η γνωμοδότηση για τη συνεδρίαση της 8 η Μαΐου. Οπότε θα ξεκινήσει ε, να τρέχει η, τροπολογία, ε, η προθεσμία για τις τροπολογίες. Θα ψηφίσουμε στις 31 Μαΐου ε, και θα λήξει στις 31 Μαΐου και θα ψηφίσουμε τον Ιούνιο στην Επιτροπή. Okay, thank you very much Σας ευχαριστούμε πολύ, λέει ο κ. Σταυρακάκης. Ο πρώτος, ή μάλλον η πρώτη σκιώδηση συγκίτρια... Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία συντάκτρια Μαρία Ιρίκογεν Πέρες για το έργο της και να πω ότι συμφωνώ μαζί της στα περισσότερα θέματα. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα θέματα και για την Επιτροπή μας, την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, αλλά είναι πολύ σημαντικά και για τους δικαιούχους των κονδυλίων των κοινωνικών ταμείων γιατί πολλοί θα ωφεληθούν από την υλοποίηση των στόχων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Θα ήθελα να πω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ε, είναι σημαντικό εργαλείο για την καταπολέμηση της ανεργίας, της καταπολέμησης της φτώχειας, του περιορισμού των κοινωνικών ανισοτήτων και θα πρέπει να μας επιτρέψει να επενδύσουμε στο ανθρώπινο δυναμικό και να προωθήσουμε τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης που θα έχουν ποιοτικό χαρακτήρα και θα είναι όσο το δυνατό περισσότερες στα πλαίσια και της στρατηγικής του 2020. Κατά τη γνώμη μου, τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου θα πρέπει να έχουν ως προτεραιότητα τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων απασχόλησης, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την πρόσβαση σε αγορά εργασίας των μακροχρόνιων έργων ε, ηλικιωμένων νέων ή γυναικών. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να είναι η προτεραιότητα για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και έτσι θα αποφέρουν καρπούς και δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν από αυτό. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική η συζήτηση για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και στα πλαίσια αυτής αναφέρεται και η ανάγκη να γίνει μια αποτίμηση της λειτουργίας και των αποτελεσμάτων από τη χρησιμοποίηση των κονδυλίων του ΕΚΤ, ώστε ναι μεν να είμαστε ικανοποιημένοι όταν υπάρχει ψηλό ποσοστό απορρόφηση και εκταμίευση, αλλά θα πρέπει να πιάνουν τόπο αυτά τα χρήματα. Θα πρέπει να αξιοποιούνται σωστά τα κονδύλια. Δηλαδή, όντω να, ε, να δημιουργούνται περισσότερε θέσει απασχόληση ποιοτικέ ή να βελτιώνεται η κατάσταση στην αγορά εργασία. Θα πρέπει να γίνεται μια αποτίμηση λοιπόν των αποτελεσμάτων. Συμφωνώ με την εισηγήτρια ότι χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ελαστικότητα σε ό,τι αφορά την κατανομή των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ε, δεν χάνουμε ευκαιρία να τονίζουμε την ανάγκη ελαστικότητας και κατά τη γνώμη μου είναι επιτακτική ανάγκη σήμερα να λάβουμε υπόψη τα ιδιαίτε, τις ιδιαίτερες ανάγκες κοινωνικές και οικονομικές των διαφόρων περιφερειών. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα κουστούμι για όλους, μια λύση που να εφαρμόζεται ανελαστικά σε όλες τις περιφέρειες, σε όλες τις χώρες, γιατί υπάρχουν μεγάλες κοινωνικές και οικονομικές διαφορές. Δεν θέλουμε άκαμπτα μοντέλα για την κατανομή των κονδύλιων του ΕΚΤ γιατί έτσι δεν θα μπορέσουμε να στηρίξουμε πραγματικά τους τομείς και τις περιφέρειες που χρήζουν παρέμβασης και ενίσχυσης. Ο προγραμματισμός των δράσεων του Κοινωνικού Ταμείου θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη αυτή τη διαφορά των αναγκών. Γι' αυτό και θα πρέπει στο άρθρο 4 το θέμα της ε, θεματικής συνοχής ε, να το φροντίσουμε ώστε να υιοθετήσουμε μια σωστή διατύπωση. Χρειάζονται κάποιες διευκρινήσεις ε, ως προς τις προτεραιότητες επίσης. Θα πρέπει να προβλέψουμε τι ακριβώς παρεμβάσεις μπορεί να χρηματοδοτήσει το κοινωνικό ταμείο και υπό το πρίσμα και των αποτελεσμάτων. Οι δείκτες είναι πολύ σημαντικό θέμα και για την, το προγραμματισμό αλλά και για τα επιχειρησιακά προγράμματα ή το ανθρώπινο δυναμικό. Ένα άλλο σημαντικό θέμα. Πρέπει να έχουμε επάρκεια δικτών ώστε να μπορούμε να αποτιμήσουμε την αποτελεσματικότητα της χρησιμοποίησης των κονδυλίων του ΕΚΤ. θα πρέπει να κρίνουμε, ε, ως, στους δείκτες να περιλαμβάνουμε τον αριθμό των δικαιούχων, τα αποτελέσματα που ε, επιτύχαμε. Χρειάζονται λοιπόν τέτοια στατιστικά στοιχεία και να λαμβάνονται υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των επαρχιών, των περιφερειών. Δεν θα πρέπει αυτόματα να εφαρμόζονται οι δείκτες. Οι ιδιαιτερότητες θα πρέπει να λαμβάνονται ανα πάσα στιγμή υπόψη. Επίσης δεν υπάρχουν συστηματικές λύσεις ό,τι αφορά τα εκπαιδευτικά συστήματα ή τα συστήματα επαγγελματικής κατάρτισης. Ούτε δίνουμε αρκετά ε, ενάυσματα στους εργοδότες προκειμένου να πάρουν σε στάση, σε ασκήση νέους. Είναι κρίμα να μην υπάρχει κάτι τέτοιο. Αυτό το στοιχείο θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στους δείκτες αξιολόγησης ε, των προγραμμάτων, των επιχειρησιακών προγραμμάτων για το ανθρώπινο δυναμικό, για παράδειγμα, το ανθρώπινο κεφάλαιο. Περιμένουμε λοιπόν με ανυπομονησία την γνωμοδότηση της κυρίας Πέρες για την οποία θα καταθέσουμε και κάποιες τροπολογίες. Πάντως πιστεύω ότι οι τροπολογίες αυτές απλώς θα εμπλουτίσουν και θα ενισχύσουν ουσιαστικά τη γνωμοδότηση προκειμένου να γίνει καλύτερη αξιοποίηση και να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Σας ευχαριστώ κυρία Σρέντερ. <coughs> Ευχαριστώ και εγώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Συγγήτρια, το ξανακοίταξα, δεν είναι διαθέσιμη η έκθεση. Ακόμα δεν μπορούμε δηλαδή να δούμε γραπτά τα όσα μας είπατε. Όμως, σημαντικά θέματα τα οποία έχουμε συζητήσει και μαζί σας. Πρώτα, ο προγραμματισμός. Στο άρθρο 4.3 το έχει περιορίσει η Κομισιόν με τρόπο που δεν είναι δυνατόν να ενταχθεί στο πλαίσιο. Γι' αυτό έκανα μια πρόταση εγώ. Δεν νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε στις προτεραιότητες επενδύσεων. Πέφτουμε σε ένα επίπεδο των πρακτικών μέτρων αν θέλουμε και να κάνουμε, και να κάνουμε και ένα πρόγραμμα σε επίπεδο περιφέρειας, έχουμε και άλλα πράγματα, δηλαδή έχουμε 7 ή 8 ή 9 τελικά προτεραιότητες επενδύσεων μόνο για την φτώχεια, μόνο για την κοινωνική συμπερίληψη. Αν βάλω πλέον 6 από, από αυτά που λέτε εσείς, τότε δεν μπορώ να κάνω κανένα προγραμματισμό. Γι' αυτό ας προχωρήσουμε από το επίπεδο των προτεραιοτήτων επενδύσεων στο θεματικό επίπεδο που κάνει και το ΕΦΑ. Όχι αυτά τα 18, αλλά να προχωρήσουμε στο επίπεδο το θεματικό. Και να δούμε το ευρωπαϊκό στρατηγικό πλαίσιο να περιοριστεί στα σημαντικά θέματα. Είναι προφανή ποια είναι αυτά. Αναφέρονται σε αυτούς τους 11 θεματικούς στόχους. Αυτό για μένα θα σημαίνει ότι αναλαμβάνουν δέσμευση οι περιφέρειες για το ποσοστό που προτείνετε εσείς, να δώσουν τόσα χρήματα για τρία θεματικά αντικείμενα. Το κεφάλαιο δηλαδή 9 του Γενικού Κανονισμού, δηλαδή τον τομέα της απασχόλησης, της κοινωνικής συμπερίληψης και καταπολέμησης της ανεργίας, εκπαίδευσης, κατάρτισης και διαβίου κατάρτισης, να υποστηρίξουν λοιπόν αυτά. Και αυτό θα σημαίνει για τις περιφέρειες ότι θα έχουν 16 προτεραιότητες επενδύσεων με τι οποίε να μπορούν να επιτύχουν αυτού του στόχου. Έχουν λοιπόν μια ελευθερία, μια ευελιξία, όπω τη χρειάζονται πραγματικά οι περιφέρειες, για να φτάσουν στους σκόπους αυτού. Με τη μέθοδο αυτό, δηλαδή, με αυτή, αυτή, δηλαδή να περάσουμε σε αυτό το θεματικό επίπεδο, στο θεμα, στους θεματικούς στόχους δηλαδή, όπως κάνει και το ΕΦΡΕ. Τώρα, εγώ έχω υποβάλει και γραπτά μια πρόταση, την οποία θα σας διαβιβάσω ευθύ αμέσως και νομίζω ότι τα διευκρινίζει τα πράγματα αυτά που λέω. Και έχω συζητήσει και με άλλους, έχω συζητήσει και με πρόσωπα της διοίκησης και όλοι έχουν συμφωνήσει. Διότι η πρότασή μου ξεκαθαρίζει τα πράγματα, τα τοποθετεί απλά και ξεκάθαρα και στηρίζει την κοινωνική πολιτική στην Ευρώπη. Θα σας τη δώσω λοιπόν γραπτά την πρόταση αυτή. Αν την διαβάσετε νομίζω θα αντιληφθείτε καλά το νόημα. Δεύτερο, σας υποστηρίζω για την ε, αρχή της partnership, δηλαδή άρθρο 6. Εδώ δεν είναι βέβαια παρούσα η Γενική Διεύθυνση Ρέγγιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σήμερα το πρωί αντιμετώπισε βέβαια την κριτική για όλους τους στόχους της. Αλλά αν έρθω στο άρθρο 1, τι έχει κάνει εκεί η Γενική Διεύθυνση Ρέγγιο. Από τη μια μεριά βάζει στη διάθεση των ε, εταίρων ένα global grant ώστε να είναι σε θέση να συνομιλήσουν ισότιμα με τις διοικήσεις. Υπάρχει δηλαδή το, παράδειγμα της best practice, ο Γιάνν Όλσεν από την Ευρωπαϊκή και Κοινωνική Επιτροπή το εξήγησε, εκεί δηλαδή όπου οι εταίροι έχουν ένα μικρό γραφείο το οποίο τους υποστηρίζει στην προπαρασκευή για να μπορούν να συζητήσουν όπως είπα ισότιμα με τις ε, ε, διοικητικές αρχές, τότε εκεί λειτουργεί το σύστημα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό το κατανόησε η Κομισιόν και έχει φτιάξει ένα είδος global grant, μιας ε, σφαιρικής ας πούμε επιχορήγησης. Έχει καλός λοιπόν εδώ. Μετά όμως τι προτείνει. Λέει αυτό το grant θα χρηματοδοτείται από τους διάφορους άξονες προτεραιοτήτων. Αυτό σημαίνει ότι οι εταίροι θα πρέπει να πάνε σε κάθε άξονα προτεραιότητας και να πούν σας παρακαλώ δώστε μας λίγο λεφτά για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε λίγο το γραφείο μας και να μπορέσουμε να μπορούμε να συνομιλούμε, να μπορέσουμε να συνομιλούμε με, την, ε, με τη διοίκηση ισότιμα. Αυτό όμως είναι καταδικασμένο σε αποτυχία εξ αρχής και γι' αυτό θα ήθελα να διαγράψω την ιδέα αυτή. Αν ήταν εδώ εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Ρέγγιο πάλι θα θύμωνε διότι θα του είχαμε διαγράψει άλλη μια ιδέα. Αλλά δεν είναι δυνατόν να απαιτήσουμε από μια μη κρατική οργάνωση να σηκωθεί να πάει σε 10 διαφορετικέ υπηρεσίε στην χώρα μέλο και να λέει σα παρακαλώ δώστε μου λίγα λεφτά εσεί, εσεί, εσεί για να μπορέσω να κάνω μια δουλειά την οποία κάνω εθελοντικά και η οποία έχει μια κοινωνική προστιθέμενη αξία, επειδή εμεί οι Ευρωβουλευτέ θεωρούμε ότι είναι σημαντικό. Τώρα, θα πρέπει να του διευκολύνουμε το έργο αυτό Γι' αυτό εδώ πρέπει να κάνουμε μια μικρή διαγραφή. Βέβαια θα θυμώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως είπα και πριν, αλλά δεν υπάρχει και άλλος τρόπος. Το τελευταίο που είναι σημαντικό για μένα, εν προκειμένου, είναι το ζήτημα των δικτών. Μπαίνουμε εδώ τώρα νομίζω σε μια ευρύτερη συζήτηση. Είναι η συζήτηση δηλαδή που κάναμε και με τον Γιάνν Ολβριχτ στο ΕΦΡΕ. Δηλαδή για τη συνολική αντίληψη και εκεί είναι διαφορετικές οι απόψεις, οι απόψεις που προβάλλουν οι κύριοι Βαν Ρόι και Κρέλ. Πρέπει να συνομιλήσουμε στην ομάδα εργασίας ποια δομή θα δώσουμε, πώς θα γίνει η επίδοση, ποια μορφή θα έχει η performance δηλαδή, ποιους δείκτες θα επιλέξουμε. Από την άλλη μεριά, είναι απαραίτητο να πάμε και στο επίπεδο του νομοθετικού, το νομοθετικό, δηλαδή τον κανονισμό. Όμως τότε οι δείκτες γίνονται πολύ τυπικοί και δεν έχουν πολύ ουσιαστικό περιεχόμενο. Αν πούμε δηλαδή οι άνθρωποι από την τάδη ηλικία μέχρι την τάδη ηλικία, για παράδειγμα 64, που έχουν λάβει, που έχουν απασχόληση. Αυτός είναι ένας δείκτης. Αλλά έχουν πάρει μια δουλειά, έχουν δηλαδή βρει μια απασχόληση από την οποία να μπορούν να ζήσουν ή παρόλη την απασχόληση αυτή πάνε και ζητάνε και κοινωνική στήριξη, δηλαδή ε, ε, λεφτά από την κοινωνική ασφάλεια. Επίσης η σύμβαση που πέτυχαν μήπως διαρκεί ένα δίμηνο και μετά λίγη ή είναι επίπεδου κατώτατου ημερομισθίου κλπ. Επομένως δεν λέει αυτό τίποτα εάν έχουμε πράγματι επιτύχει τον στόχο της απασχόλησης. Και γι' αυτό πρέπει να καθίσουμε να σκεφτούμε τι θα κάνουμε με τους διάφορους δείκτες. Ο Γιάνν Όλμπριχτ είναι πάντοτε πιο μπροστά από όλου μα, τρία βήματα πιο μπροστά και έχει κατανοήσει που κολλάει το θέμα. Υπάρχουν διάφοροι δείκτες, ορισμένοι δείκτες υπάρχουν για να μπορέσω να ξαναπάρω τα χρήματά μου και θα πρέπει να είναι στο χαμηλότερο, στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο. Υπάρχουν βέβαια και οι δείκτες έκροων που έχουν νόημα γιατί δεν μπορώ ως διοίκηση να εξασφαλίσω ότι θα γνωρίζω ποιος έχει απασχόληση και ποιο καιρό. Αλλά τον έχω εκπαιδεύσει, το έχω εκπαιδεύσει το συγκεκριμένο άτομο και έχω δικαίωμα να ξαναπάρω τα λεφτά μου πίσω. Αυτό πρέπει να το σκεφτούμε όταν θα γράφουμε τον κανονισμό. Αλλά υπάρχουν και άλλοι δείκτες που δεν λειτουργούν. Και γι' αυτό πρέπει να κάνουμε τη συζήτηση αυτή. Και αν δώσουμε τώρα νομοθετικό χαρακτήρα στους δείκτες αυτούς, πρέπει να το σκεφτούμε, διότι χωνόμαστε σε ένα στενό κορσέ. Και αυτοί οι οποίοι τελικά θα χρησιμοποιήσουν τα χρήματα αυτά, μπαίνουν και αυτοί στον στενό κορσέ. Θα μπορέσουν εν τέλει με τον κορσέ αυτό να πετύχουν αυτά που θέλουμε να πετύχουν. Εγώ είμαι υπέρμαχος να πετύχουν τους στόχους της Ευρώπης 2020 ή τα διαφθορτικά ταμεία. Αλλά δεν νομίζω ότι όλα αυτά τα κορσέ βοηθάνε να το πετύχουμε αυτό. Σκέφτομαι λοιπόν εσάς, Λάμπερτ, άξονες προτεραιότητες, common strategy framework και δείκτες, όλα αυτά, εάν τα βάλετε στο νομοθετικό επίπεδο, δεν ξέρω. Έχω λοιπόν τις επιφυλάξεις μου μήπως δεν εξυπηρετούμε το σκοπό. Δηλαδή μήπως τα έρουμε σε ένα τέτοιο υψηλό επίπεδο που τελικά είναι ακόμα πιο στενό ο κορσές. Αυτό λέω και εν τέλει λέω να τα συζητήσουμε όλα αυτά ανοιχτά. Ευχαριστώ. Κύριε Βανίστρη Ροϊ. Uh, uh, Ευχαριστώ πολύ. Ιδιαίτερα για την βαθύτατη ανάλυση την οποία μόλις ακούσαμε και για τη συνεισφορά φυσικά της εισηγήτριας αυτή την προσπάθεια που κάνατε να τη και σε εμά, όχι μόνο στην εισηγήτρια, γιατί θα μας βοηθήσει. Γνωρίζω ότι είσαστε και προσωπικά επίσης δραστηρία στην Επιτροπή Απασχόλησης. Οπότε πρέπει να δώσετε και εκεί ένα σκληρό αγώνα και όπως είπατε θα πρέπει να ισχύσει η ίδια λογική και στις δύο κοινοβουλευτικές επιτροπές. Είναι λίγο περίεργο να βλέπει κανείς ότι οι χώρες θα αποφασίζουν σε ποιο επίπεδο θα χρησιμοποιούν το περιφερειακό και το κοινωνικό ταμείο. Αν θέλουμε να υπάρξει πραγματική συνέργεια όλων των εμπλεκομένων, θα πρέπει να υπάρχει θα έλεγα μια αναλογία στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα ταμεία αυτά. Αν υπάρχουν διαφορετικού τρόπου χρήσης και διαφορετικά ταμεία που χρησιμοποιούνται σε κάθε χώρα για την επίτευξη αναλόγων στόχων, δημιουργείται ένα πρόβλημα. Πώς θα μπορέσουμε να πούμε στις πόλεις σαν παράδειγμα πώς μπορούμε να εξηγήσουμε στις πόλεις, στις αστικές περιοχές, ε, με ποια μέσα θα επιδιώξουν να πετύχουν τους στόχους τους οποίους έχουν θέσει, όταν πρέπει κάθε φορά να χρησιμοποιούν διαφορετικά επίπεδα επεξεργασίας, παρουσίασης προγραμμάτων και χρηματοδότησης τελικά. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει ε, μια ισοτιμία στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα διαθέσιμα μέσα και σαν παράδειγμα έχω τις ε, συμβάσεις εταιρική φύσης. Η Επιτροπή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν μπορώ να σχολιάσω τις τροπολογίες γιατί δεν τις έχουμε δει ακόμα. Κάποιες από αυτές δείχνουν πάντως ότι θα μας βοηθήσουν να ξεκαθαρίσουμε τον κανονισμό και να τον κάνουμε πιο αποφασιστικό που αυτό χρειάζεται. Περιμένουμε λοιπόν να λάβουμε το κείμενο από την εισηγήτρια, ιδιαίτερα σχετικά με την ενίσχυση της ισότητας των φύλων και την εμπλοκή όλων των ενδιαφερομένων. Το πρόγραμμα αυτά τρόφιμα για τους περισσότερο φτωχούς για τους περισσότερο απόρους. Ξέρετε τι έγινε η συζήτηση την προηγούμενη ολομέλεια στο Στρασβούργο. Η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκμεταλλευτεί τη δυνατότητα πρωτοβουλία την οποία έχει και θα επανέλθει με μια συγκεκριμένη πρόταση για τη συνέχιση του προγράμματος αυτού αλλά με ένα διαφορετικό τρόπο. Θα έχετε πληροφορίες μετά τις καλοκαιρινές διακοπές αλλά όχι αυστηρά μέσα από το ε, κοινωνικό ταμείο. κάποια επιπλέον σχόλια τα οποία χρήζουν διευκρινήσεων. Για τους δείκτες. Ίσως να επαναλάβουμε εδώ ότι οι δείκτες τους οποίους έχουμε προτείνει για όλα τα ταμεία είναι ε, οι ελάχιστοι κοινοί δείκτες. Εμείς πιστεύουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε τη συμφωνία με τα κράτη-μέλη σχετικά με την ε, υποχρεωτική χρήση τους. Προφανώς και θα πρέπει να υπάρξουν κάποιοι ειδικοί δείκτες οι οποίοι να ξεπερνούν το κοινό πλαίσιο το οποίο έχουμε εμείς και στο κοινωνικό και στο περιφερειακό ταμείο. Αλλά από την άλλη δεν νομίζω ότι μπορούμε ε, να συμφωνήσουμε με περισσότερους δείκτες και όταν λέω να συμφωνήσουμε να υπάρξει μια συμφωνία κοινός παρανομαστής Κρατάμε λοιπόν ορισμένους δείκτες οι οποίοι μας επιτρέπουν να σας μεταφέρουμε τα συνολικά επιτεύγματα των ταμείων, ταμείο και ταυτόχρονα να υπάρχει η δυνατότητα ε, να μπορούμε ε, σε εθνικό ή σε περιφερειακό επίπεδο να σας μεταφέρουμε στοιχεία. Σχετικά με τους μηχανισμούς συγκέντρωσης, εμείς έχουμε ήδη εξηγήσει ότι οι μηχανισμοί τους οποίους έχουμε προτείνει για το κοινωνικό ταμείο είναι οι σωστοί θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να ζητήσουμε τα κράτη-μέλη ή τις περιφέρειες να κάνουν αυτή τη διάκριση ανάμεσα στην απασχόληση, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού ε, κτλ. Νομίζω ότι ε, σε όλους αυτούς τους τρεις στόχους μπορούμε να προχωρήσουμε και περιμένουμε βέβαια το σύνολο των προτάσεων τις οποίες θα κάνετε εσείς και ίσως προφανώς και η Επιτροπή Απασχόλησης. Τώρα για το 6.1, άρθρο 6, παράγραφος 1. Το 6.1 στην ουσία δίνει τη δυνατότητα, υπενθυμίζει ότι υπάρχει δυνατότητα για τις περιφέρειες ή για τα κράτη-μέλη να εκχωρούν την εκτέλεση τμήματων ή ολοκλήρων προγραμμάτων σε μη κυβερνητικέ οργανώσεις είναι κάτι το διαφορετικό από το ITI, αλλά είναι μια δυνατότητα εκχώρησης αρμοδιότητας η οποία δεν έχει μια εδαφική αν θέλετε δυναμική, είναι όμως ε, δυνατότητα που δίνει σε μη κυβερνητικέ οργανώσεις να διαχειριστούν τμήματα προγραμμάτων. Βέβαια αυτό θα πρέπει να διευκρινίζεται κάθε φορά ε, Ξέρουμε σαν παράδειγμα ότι ο Ερυθρός Σταυρός στο πρόγραμμα Λούτσα στην Ισπανία έχει την δυνατότητα να προχωρήσει ορισμένα θέματα καλύτερα από εμά και ε, προσπαθούμε να εκτιμήσουμε και σωστά τις θεσμικές ικανότητες σε οργανωτικό ενώ επίπεδο τις οποίες μπορεί να έχουν ορισμένες μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Τώρα, για τις επιδόσεις, την ιδέα των επιδόσεων και τον δίκτυο αυτό, αν τον αποκλείσουμε, τότε μπορούμε να αποκλείσουμε όλους τους δίκτες. Οπότε σε αυτή την περίπτωση τίθεται το θέμα αν πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι δίκτες ε, έτσι κι αλλιώ. Και αυτό το είχε πει και ο κύριος Μάρτιν. Ευχαριστώ Μαρία. Έχεις να προσθέσεις κάτι. Muchas gracias, muchas gracias, Presidenta. Agradezco... Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους. Και εγώ θέλω το συντομότερο δυνατό να ετοιμάσω την γνωμοδότηση, να μεταφραστεί. Ελπίζω την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου ήδη θα είναι έτοιμη, για να μπορέσουμε να έχουμε διάλογο ε, πιαπτών προτάσεων, γραπτών και τροπολογιών επίσης. Ευχαριστώ την κυρία Γουκασίτσευσκα για τα σχόλιά της είπα και εγώ ότι θα πρέπει το ταμείο αυτό να είναι όσο πιο αποτελεσματικό γίνεται. Και φυσικά επενδύουμε στους ανθρώπους, στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Αυτό είναι το σημαντικότερη πτυχή ε, του κοινωνικού ταμείου και φυσικά μας ενδιαφέρει και η ποιότητα της απασχόλησης. Θέλουμε να αποτιμήσουμε τα αποτελέσματα του ΕΚΤ, να δούμε τις επιτυχίες που είχε και είναι δύσκολο βέβαια να δούμε πόσες φορές μπαινοβγαίνει κάπως, από την αγορά εργασίας. Αλλά θα πρέπει να του δώσουμε τα εφόδια ώστε να μπορέσει να ανακτήσει ε, τη δουλειά του ή να βρει μια νέα θέση στην αγορά εργασίας. Ευχαριστώ την κυρία Σρέντερ για τα σχόλιά της και είμαι βεβαία ότι μόλις λάβει ένα και το κείμενο θα διαπιστώσει ότι πολλές από τις τροπολογίες μου συμβαδίζουν με τις απόψεις της. Ευχαριστώ και τον ε, κύριο Βανίστρε Ρόι Σίγουρα ε, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μια συνοχή και συνέπεια μεταξύ των ταμείων, να αποφύγουμε την επικάλυψη μεταξύ των ταμείων, ιδιαίτερα στο ΕΚΤ. Επίσης, ε, ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις πληροφορίες που μας έδωσε και περιμένουμε την πρόταση από τον Επίτροπο σε ό,τι αφορά ε, το πρόγραμμα τροφίμων για τους απόρους ε, που θα υποβληθεί πριν ή μετά το καλοκαίρι. Ευχαριστώ και μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο, το σημείο 13. Έχουμε κάποια απόφαση. Άλλε διευκρινήσει δεν χρειάζονται. Περάμε στο 13 λοιπόν, τη γνωμοδότηση τη Επιτροπή μα ό,τι αφορά την εντολή για τον τριμερή διάλογο για τον προπολογισμό του 2013. Συγκεκριτή μα ο κύριο Σταυρακάκη. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, για άλλη μια χρονιά η συζήτηση για την κατάρτιση του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιείται με την οικονομική και κοινωνική κρίση να βάζει σε δοκιμασία τους προπολογισμού όλων των χωρών. Παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι προπολογισμοί καταρτίζονται στη βάση εξορθολογισμού των δημοσιονομικών δαπανών και σκληρών οικονομικών μέτρων σε πολλού τομεί τη οικονομία. Ωστόσο, είναι απαραίτητο ο δημοσιονομικό εξορθολογισμό να εξορροπηθεί με τι κατάλληλε επενδύσει αφενός για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται από τις αιτήκες και αφετέρου για να αντισταθμιστούν οι αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η πολιτική συνοχή έχει αποδείξει την προστιθέμενη αξία της. Η πολιτική συνοχή θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως το κατάλληλο παιδιτικό μέσο που θα οδηγήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση στην ανάπτυξη και στην δημιουργία θέσεων εργασίας με το να αντιμετωπίσει με ακρίβεια τις επενδυτικές ανάγκες των περιφερειών. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα συμβάλλει μονάχα στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών, αλλά και στην οικονομική ανάκαμψη και ανάπτυξη ολόκληρη τη Ένωση. Στην γνωμοδότησή μου κάνω ιδιαίτερη μνήμα στο πρόβλημα το οποίο από το Δεκέμβριο απασχολεί την Επιτροπή Προπολογισμών. Είναι το πρόβλημα των καθυστερημένων πληρωμών. Η επιτάχυση τη υλοποίηση των περισσότερων προγραμμάτων τη πολιτική συνοχή οδήγησε στο τέλο του 2011 σε ένα σημαντικό αριθμό καθυστερημένων πληρωμών που έπρεπε να αντιμετωπιστεί μέσω της διάθεσης επαρκών πιστώσεων πληρωμών το 2012. Στις 18 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια της Επιτροπής Συνδιαλλαγής στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τον προπολογισμό του 2012, στην οποία συμμετείχα για 16 ώρες η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έγινε μάρτυρας ενός πικ-πονγκ μεταξύ Συμβουλίου και Επιτροπής σχετικά με τα ακριβή στοιχεία του προπολογισμού. Επί 16 ώρες το Συμβούλιο αφισβητούσε και η Επιτροπή αντέκρου τους χειρισμού του Συμβουλίου. Τελικά, όπως γνωρίζετε, το Συμβούλιο κατάφερε να περάσει τη γραμμή του σχετικά με ένα περιορισμένο επίπεδο πιστώσεων πληρωμών και εμείς, ως αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου, αναγκαστήκαμε να συμφωνήσουμε για να μην αβαγήσουν οι διαπραγματεύσεις. Εν προκειμένου στη γνωμοδότηση εκφράζω την ανησυχία ότι αυτές οι ελλείψεις πληρωμές είναι πιθανόν να επιδεινωθούν και το 2013, όπου η εφαρμογή των προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής αναμένεται να έχει επιταχυνθεί. Γι' αυτό το λόγο κάνω έκλειστο στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβούν με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην άμεση ανάλυση και αξιολόγηση των ποσών και των αναγκών, προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο η εφαρμογή των προγραμμάτων για το 2013. Η έλλειψη στις πιστώσεις πληρωμών θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την εύρεθμη εκτέλεση των προγραμμάτων. Επίσης, στη γνωμοδότηση γίνεται έκκληση προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αξιολογήσουν προσεκτικά τις πραγματικές ανάγκες όσο αφορά τις πληρωμές στον τίτλο 1β, να μην προβούν σε περικοπές που να είναι μη ρεαλιστικές και αβάσιμες και που να αντιβαίνουν στις προβλέψεις που παρέχουν τα ίδια τα κράτη-μέλη, οι οποίες χρησιμεύουν ως βάση για την κατάρτιση του σχεδίου προπολογισμού. Το κύριο μήνυμα της γνωμοδότησης είναι ότι σε αυτή την περίπτωση θα αντιταχθούμε σε κάθε ενδεχόμενη μείωση στο επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών σε σύγκριση με τις ανάγκες και θα εκτιμηθούν από την Επιτροπή στη βάση αυτή. Τέλος, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η προθεσμία για να υποβάλλετε τις προτάσεις σας στη Γραμματεία σχετικά με τα πιλωτικά σχέδια και τις προπαρασκευαστικές δράσεις που προτείνει η Επιτροπή μας είναι στις 11 Μαΐου. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω κανένα σκιώδη γιατί στην αίθουσα. Θέλει άλλος κανείς το λόγο. Ο Φρανσουά Αλφόνση. Σας είχα μπροστά και δεν σας έβλεπα. Θα ήθελα να πω στον κύριο Σταυρακάκη ότι συμφωνώ με τη γνωμοδότηση, σωστά εντοπίζει τις προτεραιότητες και η συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2013 δίνει τις βασικές κατευθύνσεις και για τη συζήτηση που θα έχουμε για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το MFF. Λυπούμε, έχουμε κουραστεί όλοι. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι θα πρέπει να υιοθετήσουμε μια στεναρή θέση ότι η περιφερειακή ανάπτυξη, το, το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής μας επιτρέπουν να αντιμετωπίσουμε με αποτελεσματικό τρόπο την κρίση. Οι δράσεις του ε, Ταμείου Συνοχής είναι αντικυκλικές, δηλαδή βοηθά το Ταμείο Συνοχής στις ε, πιο μειονεκτικές περιοχές να ξεπεράσουν τις δυσκολίες με δεδομένες διαδικασίες και γνωστές και με τρόπο που να εξυπηρετούν το κοινό συμφέρον της Ευρώπης. Και η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της κρίσης έγκυται στην ενίσχυση της πολιτικής συνοχής. Πιστεύω ότι αυτό το πολιτικό διάβημα ε, αναφέρεται και εντοπίζεται πολύ σωστά στη γνωμοδότηση και περισσότερο από ποτέ είναι ανάγκη να διατρανώσουμε αυτή την ε, θέση ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε την ε, πολιτική συνοχή, πολλά δε μάλλον που η χρηματοδότησή τη πολλέ φορέ αφισβητείται στι μέρε μα. Αν δεν θέλει άλλο κανεί το λόγο, δεν ξέρω κύριε Σταυρακάκη αν θέλετε να επανέλθετε. Thank you very much. Ε, ε θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Φρεσουάλ Φώση για τις παρατηρήσεις του και ελπίζω ότι με τη συνεργασία μα και τι τροπολογίε που ενδεχομένω θα καταθέσουν οι συνάδελφοι θα μπορέσουμε να συνεισφέρουμε στο σχηματισμό μια ενιαία και δυνατή διαπραγματευτική θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον επερχόμενο τρίλογο επί τη σχεδίου του προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2013. Thank you. Thank you. Σας ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε... Α, με συγχωρείτε. Ναι, ναι, η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών. 3η Μαΐου το μεσημέρι, το μεσημέρι στις 12. 14 τώρα. Γνωμοδότηση του κυρίου Ολέζνιτσακ. Διευρωπαϊκές Ενεργειακές Υποδομές. Ευχαριστώ. Η γνωμοδότησή μας καθορίζει τα κριτήρια για τα διευρωπαϊκά δικτύα των ενεργειακών υποδομών που θα αποτελέσουν το αντικείμενο ε, κοινού ενδιαφέροντος, συστηματοποίηση της εφαρμογής και της παρακολούθησης ε, του σχεδίου, η εξασφάλιση της ε, ανάμειξης των πολιτών και η σωστή αδειοδότηση, καθώς και οι βάσεις για τα σχέδια αυτά, επιτρέπει τη χρηματοδότηση τέτοιων διασυνοριακών προγραμμάτων. Επίσης, ο κανονισμός μιλάει για 20 προτεραιότητες και διαδρόμους και κατηγορίες διαδικασιών για χρηματοδότηση. Η πρόταση είναι καλό βήμα προκειμένου να περιοριστεί ο χρόνος αδειοδότησης για την δημιουργία σημαντικών ενεργειακών υποδομών. Έχουμε μεταξύ 10 και 12 χρόνια. Θέλουμε αυτό το διάστημα να το μειώσουμε στα 2 με 3 χρόνια για τη χορήγηση άδεια. Ε, επίσης θα πρέπει να ε, μπορέσουμε να μοιραζόμαστε όχι μόνο τα κέρδη, ε, να μην αναλαμβάνουμε μόνο κοινωνικά τις ευθύνες, αλλά να μοιραζόμαστε και τα κέρδη. Γι' αυτό και θα πρέπει να αναλαμβάνονται κάποιες ε, αποφάσεις για την αυτοχρηματοδότηση κάποιων διευρωπαϊκών και διασυνοριακών ενεργειακών σχεδίων. Οι τροπολογίες μου στόχο έχουν την εξορρόπηση των κριτηρίων των διαφόρων σχεδίων που αποτελούν ε, σχέδια κοινού ενδιαφέροντος και θέλω να επικεντρωθώ στην μεγαλύτερη δυνατή αποδοτημότητα των σχεδίων και να συγχρηματοδοτούν αυτά που έχουν ε, θετικά, ε, θετικές επιπτώσεις και εξυπηρετούν το κοινό συμφέρον. Σε ό,τι αφορά το τομέα του φυσικού αερίου, είναι πολύ σημαντικό το φυσικό αέριο και για τις περιφέρειες, γι' αυτό και χρειαζόμαστε ένα κατάλογο τέτοιων σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος και προτείνω ένα, μια διασταλτική ερμηνεία της υποδομής φυσικού αερίου, ώστε να περιλαμβάνει και τους ε, και τι εγκαταστάσει υγροποιημένου φυσικού αερίου, τι υπόγειε αποθήκε και Γιατί δεν είναι βεβαιωμένο το φυσικό αέριο ανανεώσιμη πηγή ενέργεια, αλλά η χρήση του σε ευρία κλίμακα μας επιτρέπει να περιορίσουμε την καύση άνθρακα. Νομίζω ότι ε, με επιτυχημένες επενδύσεις στις ενεργειακές υποδομές ε, θα ε, έχουμε πολύ θετικά αποτελέσματα αρκεί να μειώσουμε και τις διατυπώσεις και τη γραφειοκρατία. Η αρμόδια για καθήλη για την έκθεση αυτή είναι η Επιτροπή Ήτρε. Ευχαριστώ εκ μέρους του ΕΛΚ. Η συγκέντρη είναι η κυρία Κολάρσκα Μπομπίνσκα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Λένιτσακ για την γνωμοδότηση αυτή. Και εγώ συμφωνώ ότι το αρχικό κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πολύ καλό και οι τροπολογίες του συντάκτη της επίση επίσης είναι σωστές και νομίζω ότι θα τύχουν υποστήριξη από όλες τις πολιτικές παρατάξεις. Θα ήθελα να επισημάνω δύο ζητήματα που κατά τη γνώμη μου είναι σημαντικά. Καταρχήν, είναι αμφίβολος κάπως ε, και δημιουργεί προβληματισμό τρόπος ε, λήψης απόφασης στις περιφερειακές ομάδες για την ε, επιλογή των προγραμμάτων. Οι οργανωτές των προγραμμάτων όταν ανήκουν σε ομάδε αυτές δεν θα πρέπει να έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν το λόγο σε τέτοιες αποφάσεις. Αυτό λέει ο συντάκτης ε, και τη έκθεση ΙΤΡΕ, το τόνισε και ο συντάκτης τη δικής μας γνωμοδότησης, γιατί ε, αν ο οργανωτής του προγράμματος συμμετέχει στην απόφαση για το δικό του πρόγραμμα, για πρόγραμμα που τον ενδιαφέρει, δημιουργείται σύγκρουση συμφερόντων. Θα πρέπει να το τονίσουμε. Επίσης, σημαντικό είναι να περιοριστούν οι καθυστερήσεις και να επιταχυνθεί η διαδικασία προκήρυξης διαγωνισμών. Το θέμα είναι ποιος θα προκυρήσει τους διαγωνισμούς και ποιος θα αποφασίζει για τα αποτελέσματα των διαγωνισμών. Το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, υιοθετεί μια πιο γενική προσέγγιση και δεν περιλαμβάνει διευκρινήσεις για τα χαρακτηριστικά του διαγωνισμού και ποιες προϋποθέσεις θα πρέπει να συντρέχουν από τους υποψηφίους ε, και να πληρούνται από τους υποψηφίους. Νομίζω ότι το κείμενο θα μπορούσε να συμπληρωθεί με τέτοιες διευκρινήσεις. Και από αυτή την άποψη συμφωνώ με την πρόταση του Συμβουλίου. Θεωρώ πάντως ότι δεν είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα, είναι αυτή που θα πρέπει να οργανώνει τους διαγωνισμούς, αλλά η αρμόδιες αρχές που είναι καλύτερα εξοικειωμένες με τις ιδιαιτερότητες και τις τοπικές ανάγκες. Θα υποβάλω τροπολογίες για τα δύο αυτά θέματα και ίσως καταθέσω και μία άλλη τροπολογία που αφορά την ανταλλαγή ε, πληροφοριών με τοπικές κοινότητες. Οι υπόλοιπε τροπολογίες που θα καταθέσω είναι συντακτικού χαρακτήρα, τεχνικής φύσης, Πάντως, επαναλαμβάνω, είναι πολύ καλή η γνωμοδότηση και καλό θα ήταν να την εγκρίνουμε το συντομότερο δυνατό. Ευχαριστώ και τον εισηγητή για την αγαστή συνεργασία που είχαμε. Από ό,τι βλέπω, απουσιάζει ο Μιχάλ Τόιρερ και η Καρή Μανταλή, οπότε δεν έχουμε άλλους και οδησηγητές. Θέλει ο κανείς το λόγο για την έκθεση του κ. Λέινιτσακ. Οπότε δεν ξέρω αν κύριε Ολένιτσακ θέλετε το λόγο για να απαντήσετε. Ή μάλλον δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακαλώ, αν υπάρχει κάποιος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, thank you very much, ε, Mr. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή για τα σχόλιά του. Πράγματι η έκθεσή σας περιλαμβάνει πάρα πολλά θετικά σημεία και με τα περισσότερα από αυτά τα οποία ε, γράφετε δεν μπορούμε παρά να συμφωνήσουμε, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Δεν θα αναφερθώ στις τροπολογίες με τις οποίες συμφωνούμε, θα αναφερθώ όμως στα θέματα τα οποία μπορεί να έχουμε κάποιες διαφωνίες και δεν είναι όμως πολλά. σχετικά με την τροπολογία 6 που προσθέτει στα κριτήρια προτεραιότητας. Να πούμε εδώ ότι εμείς στα πλαίσια των κριτηρίων αυτών συμπεριλαμβάνουμε την ενέργεια και τους στόχους για την κλιματολογική πολιτική και θα πρέπει τα κριτήρια αυτά νομίζω να τα κρατήσουμε στα πλαίσια αυτών των δύο πολιτικών στόχων και να γίνει και αναφορά στα παραρτήματα για τον τρόπο καταμέτρησης των δικτών αυτών, των στόχων αυτών. Για την τροπολογία 13. σχετικά με τις ε, εγγυήσει ε, και τα δάνεια, όπως επίσης και τα δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στον τομέα των οικοδομών. Αυτό είναι κάτι το θετικό και πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα αυξήσει τις επενδύσεις της και στον τομέα της ενέργειας. Νομίζω ότι όμως η σωστή θέση για μια τέτοια τροπολογία δεν είναι κάτι το οποίο περιλαμβάνεται, μπορεί να περιληφθεί στην, στον δικό μας κανονισμό. Νομίζω ότι στο άρθρο 15 γίνεται αναφορά στα χρηματοδοτικά μέσα τα οποία μπορούν να βελτιώσουν τη ρεστότητα όπως επίσης και τη χρηματοδότηση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και από πλευράς των υπολείπων Ευρωπαϊκών Τραπεζών αλλά και της Connecting Europe, της πρωτοβουλίας του μέσου Connecting Europe. Για την τροπολογία 16. σχετικά με το να γίνει θέμα επιλογής ε, ο υπολογισμός του διαμεθοριακού κόστους, του επιπλέον κόστους στα πλαίσια της, ε, αυτού του μέσου. Πράγματι για τις ανησυχίες σας ότι η διαδικασία αυτή είναι γραφειοκρατική και μακρόχρονη είναι ακριβώς το αντίθετο. Υπάρχει ανάγκη για την ενέργεια η οποία χρηματοδοτείται από τον ιδιωτικό τομέα μέσω φυσικά αυτών οι οποίοι έχουν την εποπτεία και νομίζουμε ότι και μέσω του προϋπολογισμού του μέσου συνδέοντας την Ευρώπη, Connecting Europe, θα πρέπει να γνωρίζουμε τι είδους έσοδα προβλέπονται από τα προγράμματα αυτά μέσω των τιμολογίων τα οποία θα εφαρμόσουν στη δεύτερη φάση. Αυτό είναι κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό πριν αποφασίσουμε για τη χρηματοδότησή του ή Και αναφέρομαι πάντα στην 16. Θα πρέπει η άποψη των εποπτικών αρχών για το ύψος της χρηματοδότησης να καθορίζεται μετά από τον καθορισμό των τιμολογίων. Κάποια επιπλέον σχόλια τώρα για τα θέματα που έθωσε η κυρία Κολάσκα Μπομπίνσκα. Κατανοώ αυτό το οποίο είπατε ότι το σύστημα ή μάλλον οι εταιρείε οι οποίες αναλαμβάνουν τη μεταφορά ε, έχουν συγκεκριμένα συμφέροντα, οπότε δεν θα πρέπει να συμμετέχουν στην επιλογή των προγραμμάτων. Φυσικά και έχουν μια θέση στις διαδικασίες αυτές και πρέπει να μας εξηγήσουν περί τίνος πρόκειται ε, και τι είναι τα ακριβώς τα προγράμματα, αλλά παρόλα αυτά δεν θα κάνουν την επιλογή για τις δημόσιες προμήθειες. Σήμερα ήδη το τρίτο πακέτο δίνει τη δυνατότητα στις ρυθμιστικές αρχές να ξεκινούν ένα διαγωνισμό για συγκεκριμένα προγράμματα. Εμείς προτείνουμε να διαβρύνουμε τη δυνατότητα αυτή και να εισάγουμε επίσης ε, ε, ένα μέσο ε, τελευταίας προσφυγής, αν έχουν ληφθεί δηλαδή όλα τα απαιτούμενα μέτρα, έχουν ξεκινήσει και εξαντληθεί όλες οι διαδικασίες, αλλά δεν έχουν ξεκινήσει τα προγράμματα, τότε σε αυτή την περίπτωση το τελευταίο μέσο είναι η δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να οργανώσει αυτή το διαγωνισμό. Σύντομα λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά για την έκθεσή σας. Έχουμε λίγες ανησυχίες σχετικά με άλλες τροπολογίες. Οι περισσότερες από τις τροπολογίες που προτείνετε είναι θετικές και τις στηρίζουμε. Ευχαριστώ. Ο εισηγητής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και την κυρία Κολάσκα Μπομπίνσκα και την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νομίζω ότι μπορούμε χάρη στη συνεργασία μας να καταλήξουμε σε μια καλή γνωμοδότηση που θα ε, βελτιώσει τη δημιουργία των υποδομών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση των ενεργειακών υποδομών διορία για τις τροπολογίες είναι η 3η Μαΐου το μεσημέρι και για αυτή τη γνωμοδότηση και περνάμε στο τελευταίο σημείο της ημέρης της διάταξης την γνωμοδότηση του κυρίου Γιένς Γκάιερ για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Έχετε το λόγο κύριε Σιγητά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειακής Αναπτύξεως για το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Ένα ταμείο που αρχικά είχε ιδρυθεί για να καταστεί σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα δημοσιονομικά μέσα που διαθέτει είναι σε θέση να φανεί αλληλέγγυη με τα πρόσωπα εκείνα που ε, λόγω διαδικασιών της παγκοσμιοποίησεως τελικά πέφτουν θύματα μαζικών απολύσεων. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ορατό εργαλείο, ένα πολύ ορατό μέτρο. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση διαθέτει ιδιαίτερο, ε, ιδιαίτερη γραμμή στον προϋπολογισμό αλλά όχι ειδικό κονδύλιο. Δηλαδή εγγράφεται ένα ανώτατο ποσό που δεν φυλάσσεται όμως για το ταμείο αυτό, αλλά λαμβάνονται κονδύλια από τον προϋπολογισμό εφόσον οι χώρες μέλη καταθέσουν αιτήσει για να πάρουν χρήματα από το ταμείο αυτό. Αυτό σημαίνει ότι κάθε μέτρο πρέπει να ακολουθείται ή μάλλον ε, κάθε μέτρο πρέπει να προηγείται ειδική απόφαση και έγκρισή της για ε, λήψη χρημάτων από τον προπολογισμό. Δεν υπάρχει δηλαδή κανένα αυτοματισμό, ούτε η Κομισιόν μπορεί να δράσει αυτόνομα. Το Κοινοβούλιο πρέπει να εγκρίνει τα μέτρα που θα βοηθήσουν εκείνου οι οποίοι τελικά έχουν πέσει θύματα των μαζικών απολύσεων. Τώρα προτείνεται η συνέχιση του Ταμείου και από την Κομισιόν. το Συμβούλιο προτιμά να το καταργήσει για το αν θα συνεχιστεί ή όχι το Ταμείο βέβαια θα διεξαχθεί πολιτική συζήτηση. Εδώ πρώτα όμως πρέπει εμείς να διευκρινίσουμε το θέμα της νομικής βάσης. Η βασική αλλαγή που βλέπω να διαγράφεται τώρα απέναντι στα όσα υπήρχαν μέχρι τώρα είναι η ομάδα εκείνων που μπορεί να υποφεληθούν από το ταμείο αυτό, ότι αυτή η ομάδα δηλαδή διευρύνεται σημαντικά. Η Κομισιόν προτείνει δηλαδή στο μέλλον να περιληφθούν και αγρότες και οι διαχειριστές, δηλαδή οι, επιχειρηματίες που ηγούνται μικρών και πάρα πολύ μικρών επιχειρήσεων. Ας το πω έτσι. Εγώ διαρωτήθηκα ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι είναι πιο ευάλωτοι είναι πρώτα-πρώτα οι ανεξάρτητοι, οι αυτοαπασχολούμενοι δηλαδή, επίσης σε δεύτερο βαθμό οι μικροί επιχειρηματίες που έχουν ένα πολύ περιορισμένο κύκλο πελατών και αν αυτός μειωθεί λόγω της παγκοσμιοποίησεως, ένας μικρός κύκλος δηλαδή προσώπων στον οποίο προσφέρουν υπηρεσίες και αυτά τα πρόσωπα απολυθούν, για παράδειγμα εφόσον ε, ε μια επιχείρηση μπορεί να συμπαρασύρει και το διαφημιστικό γραφείο ή ε, αυτόν που φτιάχνει την ιστοσελίδα ε, της επιχείρησης κλπ. Αυτή, αυτό, όλοι, όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι είναι ευάλωτοι. Οι αγρότες εξ αντιθέτου, γιατί αυτό λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ενδεχομένως μπορεί με τις συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου να υποστούν ζημία οι αγρότες. Εγώ νομίζω ότι καθήκον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι, εν προκειμένου, να περιλάβει και τις πτυχές αυτές στην διαπραγμάτευση μιας τέτοιας συμφωνίας ελευθέρου εμπορίου. Ότι δηλαδή μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην αγροτική οικονομία. Τώρα το να έρχεται το ταμείο αυτό το οποίο ούτως ή έχει περιορισμένα ε, μέσα να βοηθήσει ποτέ τα πρόσωπα αυτά στην ουσία εμβαλωματικές μπορεί να είναι μόνο οι λύσεις αυτές δηλαδή δεν μπορεί να έχει ουσιώδη ε, σημασία. Στην γνωμοδότησή μου έριξα ιδιαίτερο βάρος σε αυτή την επιχειρηματολογία και να εξετάσει υπό το πρίσμα αυτό και τα διάφορα άρθρα που μας έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα αναμένω βέβαια με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις ε, απόψεις των συναδέλφων μου. Η κυρία Σρέντερ. Από ό,τι φαίνεται ο κύκλος των προσώπων που γνωρίζουν το θέμα αυτό είναι πολύ περιορισμένος από ό,τι βλέπω εδώ. Εγώ γνωρίζω την ιστορία του Ταμείου ήμουν και σκιώδης εισηγήτρια για το πρώτο, για τον πρώτο κανονισμό, έχω μερικές θεμελιώδεις παρατηρήσεις να κάνω, γιατί γνωρίζω και από την Επιτροπή Απασχόλησης ότι εκεί η έκθεση δεν έχει καν χρονοδιάγραμμα ακόμα. Διότι υπάρχουν όμως, υπάρχουν όμως ορισμένα θεμελιώδη ερωτήματα πώς γίνεται η κατανομή αρμοδιοτήτων δηλαδή λόγω αυτή τη νέα υπόθεση όπου θα καλύψει υποτίθεται και τους αγρότες, ποια επιτροπή θα είναι αρμόδια επί τη ουσία. Ο εισηγητής δεν μπορεί να κάνει τίποτα όσο δεν έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα αυτά. Ακούγεται δηλαδή να, και το ενδεχόμενο να γίνουν δύο κανονισμοί. Η Κομισιόν όμω δεν το πολύ θέλει αυτό. Και όλα αυτά είναι ασαφή ακόμη. Γι' αυτό νομίζω ότι δεν μπορούμε ακόμα να βάλουμε προθεσμία κατάθεση τροπολογιών αφού δεν γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία. Ούτε η κυρία Χάρκιν που είναι η κυρίω η δεν το γνωρίζει. Ή αν το γνωρίζει, εν πάση περιπτώσει, ας μας το πει και εμά. Από αυτά όμως εξαρτώνται πολλά. Νομίζω ότι πρέπει να σκεφτούμε ξανά ότι γεγονός είναι ότι το Ταμείο τροφοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Μα είπατε ότι τροφοδοτείται από ολόκληρο τον προπολογισμό, αλλά όλε οι σχετικέ εκθέσει μέχρι τώρα αποδεικνύουν ότι τροφοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Εγώ πιστεύω ότι εάν πρόκειται να διατηρηθεί το Ταμείο θα πρέπει να παραμείνει εκεί που είναι, δηλαδή να, να είναι ένα ειδικό εργαλείο, ένα ad hoc εργαλείο και να συνδεθεί πολύ στενότερα με το κοινωνικό ταμείο, διότι τελικά λεφτά του κοινωνικού ταμείου είναι. Α μην πλανόμεθα από πουθενά άλλου δεν παίρνει. Με την έννοια αυτή νομίζω ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε όταν θα έχει πια αποσαφινιστεί η ε, διαδικασία. Σον Κέλλη. Ευχαριστώ. Η ώρα προχωράει, γι' αυτό θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Καταρχήν πρέπει να αποφασίσουμε. Θα συνεχιστεί η λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση. Εγώ πιστεύω πως έχει νόημα να συνεχιστεί. Γιατί αυτό το ταμείο έτυχε θερμής υποστήριξη τουλάχιστον στην αρχή. Και βοηθά όσους επλήγησαν περισσότερο από την ε, ύφεση και από την παγκοσμιοποίηση. Και τώρα έχουμε την ευκαιρία να το βελτιώσουμε. Να διδαχθούμε από τα παθήματα του παρελθόντος και να καταργήσουμε τα αντιπαραγωγικά του τμήματα, βελτιώνοντάς το. Υπάρχουν σοβαρέ αδυναμίε στο Ταμείο. είμαι σκιώδη ηγητή γιατί συμμετείχα σε τρει διαφορετικέ εφαρμογέ του Ταμείου στην εκλογική μου περιφέρεια και μόνο. Υπάρχουν λοιπόν αδυναμίε που μπορεί να διορθωθούν στο Ταμείο Παγκοσμιοποίηση, προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση. Όταν ε, πρωτοαναγγέλθηκε η σύσταση του Ταμείου, ένας εργαζόμενος που έχασε τη δουλειά του είπε ότι αυτό είναι δώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή ήταν αρχικά η εντύπωση για το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Μπορεί μετά να διαψεύθηκαν αυτές τις προσδοκίες, πάντως η αρχική πρόθεση ήταν καλή. Βέβαια υπήρχαν περιορισμοί και χρονικοί, αλλά και προβλήματα εφαρμογής από τα κράτη-μέλη. Οπότε, αν είναι να συνεχιστεί το Ταμείο Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση, θα πρέπει να καταβληθεί πολύ περισσότερη ε, προσπάθεια από τα κράτη-μέλη και πολύ καλύτερο έλεγχο τη εφαρμογή και χρησιμοποίηση των κονδυλίων. Επίση, ε, είναι σημαντικό να αναμίξουμε του κοινωνικού εταίρου, ώστε κάθε άνθρωπο, κάθε εργαζόμενο που έχει χάσει τη δουλειά του να δώσει τη γνώμη του, να γίνουν γνωστά τα προσόντα του για να μπορεί να ξαναβρει μια δουλειά. Και η μείωση από 500 σε 200 ε, ε, το κατόφλι και η συγχρηματοδότηση να αυξηθεί το ποσοστό συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν συμφωνώ με τον αποκλεισμό. Ε, μάλλον είναι αυτονόητο, αυτή, αυτονόητη πρόταση για, την, για τον αποκλεισμό των γεωργιών. Των γεωργών, συγγνώμη. Αν όμως αναμορφώσουμε όντως το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης, θα πρέπει να το αφήσουμε όσο πιο ευρύ γίνεται με ελαστικότητα. Και οι γεωργοί μέχρι στιγμής επλήγησαν, οπότε ίσως από το Ταμείο Συνοχής βρουν κάποια υποστήριξη από το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Φυσικά στόχος ε, του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση είναι να ξαναβρούν όσοι έχουν χάσει τη δουλειά τους μια θέση απασχόληση. Ακόμη και οι αυτοαπασχολούμενοι. Αυτοαπασχολούμενοι είναι και οι επιχειρηματίες και οι γεωργοί. Νομίζω ότι έτσι θα είναι περισσότερη κάλυψη του Ταμείου και θα είναι και περισσότεροι οι δικαιούχοι. Θα έλεγα να υπάρχει δυνατότητα συμπερίληψης των αυτοαπασχολούμενων και των γεωργών και να μην αποκλείσουμε ε, οριζόντια οποιαδήποτε συμπερίληψή τους μπορούμε περιπτωσιολογικά να κρίνουμε αν θα συμπεριληφθεί κάποιο γεωργό ή όχι. Να μην αποκλείουμε όμω ηλίδιν του γεωργού από το πεδίο εφαρμογή. Επαναλαμβάνω, θα πρέπει να βρούμε να, να διορθώσουμε τις αδυναμίες και ω προς, το χρονικό περιορισμό, αλλά και ω προς την εφαρμογή που χώρανε σε πολλές περιπτώσει. ευχαριστώ. Όταν λέει κυρία Σρέντερ ότι οι αρμόδιες επί επιτροπές δεν έχουν προχωρήσει ακόμα αρκετά, ότι ακόμα δεν έχουν συμφωνήσει σχετικά με τις αρμοδιότητες και ποιο τμήμα θα αναλάβει πια, τότε τόσο περισσότερο είμαι ευγνώμων στον εισηγητή μας που έρχεται και μας επισημαίνει ορισμένα πράγματα που πρέπει οπωσδήποτε να προσεχθούν. Όλοι γνωρίζουμε ότι το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης ιδρύθηκε σαν εικονικό ταμείο περισσότερο για να μπορεί να απαλύνει τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης σε ορισμένες θυγόμενες περιφέρειες και να δημιουργεί κάποιες δυνατότητες απασχόλησης. Ωστόσο, κανένας ακόμα δεν έχει ορίσει τι σημαίνει επίπτωση της παγκοσμιοποίησης σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Επειδή τώρα γίνονται κάποιες προσπάθειες να περιληφθούν και οι ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην γεωργία ε, συμφωνιών ελευθέρων ε, συναλλαγών αρχίζω πλέον και δεν καταλαβαίνω καθόλου. Δεν έχω καμία κατανόηση για ε, τέτοια πράγματα. Από την άλλη μεριά είμαι υπέρ της ιδέας όπου υπάρχουν ε, βιομηχανικοί κλάδοι που είχαν κάποιο μονοπόλιο σε περιφέρειες μεγάλες και όπου τώρα ε, πάβουν να υπάρχουν διότι είναι τόσο μεγάλη πίεση της παγκοσμιοποίησης εκεί έχει καλώς προεβδομάδων λάβαμε μια απόφαση εδώ στην Ευρωβουλή που έλεγε ότι οι εργαζόμενοι της επιχείρησης Renault στη Γαλλία που χάσανε τη δουλειά τους στη Γαλλία λόγω της πολιτικής της εταιρείας διότι η εταιρεία μετέφερε την παραγωγή στην Βραζιλία και στην ε, Ασία εγκρίναμε να συμβάλλει το Ταμείο στην ανάληψη των κοινωνικών βαρών που ήταν κανονικά υπόθεση του γαλλικού κράτους και δεν έχω πάλι εδώ καμία κατανόηση γιατί πρέπει να γίνει αυτό με χρήματα του συνόλου των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Νομίζω λοιπόν πρέπει να σταθούμε κριτικά απέναντι στις μέχρι τώρα διαδικασίες που ακολουθήθηκαν και εγώ τάσομαι μάλλον υπέρ της κατάργησης του ταμείου αυτού. Άλλωστε και άλλοι λένε το ίδιο. Συχνά άλλωστε οι αιτίε είναι άλλε εκτό τη παγκοσμιοποίηση. Η πρόεδρο. Θέλετε και εσεί. Άλλοι δεν έχουν ζητήσει το λόγο. Α ε, λάβει πάλι το λόγο λοιπόν ο Γιέν Γκάιερ. Η Κομισιόν. I'm sorry, yes, εσείς, η κυρία Ιζαπέλ Πραντζίνσκι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι που ακούω αυτή τη συζήτηση εδώ. να ακολουθεί συγκεκριμένε πολιτικέ και τεχνικέ γραμμέ, οι οποίε συνολικά υποστηρίζουν το Ταμείο αυτό για το μέλλον from the implementation of the EGF in the previous phase. Έχουμε μάθει πολλά από την εφαρμογή του Ταμείου αυτού από το παρελθόν. Είχαμε συναντήσεις των ενδιαφερομένων, είχαμε συναντήσεις με τους κοινωνικούς εταίρους, είχαμε συναντήσεις με τους βουλευτές που ενδιαφέρθηκαν γι' αυτό και προσπαθήσαμε να βγάλουμε τα συμπεράσματα από τις επαφές αυτές για να βελτιώσουμε τον κανονισμό. Τελικά αποφασίσαμε να προτείνουμε τους γεωργούς γιατί και αυτοί υποφέρουν από τις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης και γιατί οι περισσότεροι από αυτούς είναι αυτοαπασχολούμενοι και σύμφωνα με τους υπάρχοντες κανονισμούς δεν μπορούσαν να πάρουν μέρος μέχρι τώρα. Δεν θα πρέπει να περιμένουμε βέβαια να εγκαταλείψουν την αγροτική δραστηριότητα και να βρουν μια νέα απασχόληση, αλλά θέλουμε να τους βοηθήσουμε να παραμείνουν ε, στην Ήπεθρο αλλά να ε, προσαρμόσουν τις δραστηριότητές τους. Δεν είναι αλήθεια ότι το Συμβούλιο αποφάσισε ότι το Ταμείο αυτό δεν θα συνεχιστεί στο μέλλον. Αυτό που συνέβη είναι ότι συζήτησε το Συμβούλιο τα θέματα, ζητήθηκε η γνώμη του και για τις αποκλήσεις κρίσεως που είχαν εγκριθεί, αν θα πρέπει να επιτρέπουμε αιτήσει για συμμετοχή στα πλαίσια της υπάρχουσας οικονομικής κρίσης και υπήρξε μία μειοψηφία η οποία μπλόκαρε το Συμβούλιο και δεν ελήφθη καμία απόφαση. Και αυτές οι αποκλήσεις οι οποίες ήταν επιτρεπόμενες μέχρι το τέλος του προηγούμενου χρόνου τώρα πια δεν υπάρχουν. Απλά. Το Συμβούλιο από την άλλη έχει μόλις ξεκινήσει τις συζητήσεις αυτές. Έχουμε εξετάσει τα άρθρα 1 με 7, την επόμενη εβδομάδα θα συναντήσουμε τα υπόλοιπα άρθρα και τα αντιμετωπίζουμε με το Συμβούλιο σε ένα τεχνικό καταρχάς επίπεδο. Δεν υπάρχει πολιτική συζήτηση σε αυτή τη φάση αν θα πρέπει να συνακιστεί το Ταμείο, αλλά μία απλή τεχνική συνάντηση. Συζήτηση, συγγνώμη. Η πολιτική συζήτηση γίνεται σε άλλα φόρα και νομίζω ότι στο τέλος το ταμείο αυτό θα είναι ένα κομμάτι του κοινωνικού ταμείου και θα μπορέσει να συνεχίσει να λειτουργεί. σχετικά με τη διεύρυνση του πεδίου λειτουργίας του. Εκτός από τις ομάδες τις οποίες ανέφερε ο κ. Γκάγερ έχουμε και εποχιακούς απασχολούμενους προσθέσει γιατί πάρα πολλοί εργαζόμενοι είναι εποχιακοί πλέον με τις επιχειρήσεις οι οποίες τους απολύουν. Έχουμε συνεργαστεί με τις εταιρείες αυτές, αλλά όταν τελειώσουν οι συμβάσεις τους οι απασχολούμενοι αυτοί δεν έχουν πλέον δουλειά, αλλά θα θέλαμε όπως έχουν ζητήσει και οι ενδιαφερόμενοι εταίροι να τους συμπεριλάβουμε στο μέλλον. Το ταμείο αυτό χρηματοδοτείται κυρίως όπως είπατε από το κοινωνικό ταμείο. Δεν είναι έτσι. Η, η διοργανική συμφωνία διευκρινίζει ότι τα ταμεία τα οποία έχουν περάσει για το ταμείο αυτό στο αποθεματικό δεν πρέπει να προέρχονται από τα διαφθρωτικά ταμεία και φυσικά όχι και από το κοινωνικό. Στο παρελθόν βέβαια ήμασταν ικανοί ορισμένες πιστώσεις πληρωμών να τις πάρουμε από ταμεία τα οποία είχαν υποχρησιμοποιηθεί και είχε χρησιμεύσει και το κοινωνικό ταμείο. Δεν συμβαίνει όμως κάτι τέτοιο. Οφελούμεθα και από το ότι το Κοινοβούλιο αποφάσισε να βάλει τις πιστώσεις πληρωμών απευθεία στη γραμμή του προϋπολογισμού μας, οπότε δεν μπορούμε να πάρουμε χρήματα αλλού, από αλλού και από την άλλη περιμένουμε να γίνει στο δεύτερο ήμιση του χρόνου η συνολική μεταφορά όταν τα χρήματα γίνουν διαθέσιμα από πολλές γραμμές του προϋπολογισμού στις οποίες υπάρχει υποχρη... υποχρησιμοποίηση. Προσπαθούμε λοιπόν να αυτοχρηματοδοτηθούμε, αλλά δυστυχώς η διοργανική συμφωνία δεν καθιστά πιστώσεις πληρωμών απευθείας διαθέσιμες για το Ταμείο, αλλά ζητά τις πιστώσεις πληρωμών να προέρχονται από ταμεία στα οποία υπάρχει υποχρησιμοποίηση. Ο κύριος Κέλλη αναφέρθηκε επίσης στο ότι ένα τμήμα του προβλήματος του Ταμείου είναι τα κράτη-μέλη, ε, είναι αυτά τα οποία δέχονται τις αιτήσει. Εμείς μέσω του Ταμείου δίνουμε στα κράτη-μέλη δύο εβδομάδες επιπλέον για να προετοιμάζουν τις αιτήσει αυτές και να είναι πλήρης οι αιτήσει έτσι ώστε η Επιτροπή στο μέλλον να μην ζητά περισσότερες συμπληρωματικές πληροφορίες από τα κράτη-μέλη, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις. Οι αιτήσει θα πρέπει να είναι πλήρης όταν κατατίθενται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αποφασίζει πολύ πιο γρήγορα από ό,τι στο παρελθόν. Ο κύριος Τζέλα είπε τι είναι η παγκοσμιοποίηση. Πράγματι ο κανονισμός περιλαμβάνει ένα ορισμό της παγκοσμιοποίησης που πολύ μας χρησιμεύσε στο παρελθόν. Τον έχουμε παρουσιάσει και στο Κοινοβούλιο όταν είχαμε αντίστοιχες περιπτώσεις και είπαμε εμείς ποια είναι τα κριτήρια της παγκοσμιοποίησης τα οποία χρησιμοποιούμε. Τώρα για το αν τα χρήματα αυτά μπορούν να ωφελήσουν μια επιχείρηση. Όχι, γιατί οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες και από την εθνική και από την κοινοτική νομοθεσία να πάρουν τα απαιτούμενα μέτρα και το έχει κάνει αυτό η Ρενό, είναι ένα παράδειγμα το οποίο δόθηκε. Ελέγχουμε το ότι οι επιχειρήσεις φέρουν εις πέρα στις υποχρεώσεις τους, αναλαμβάνουν συγγνώμη τις υποχρεώσεις τους. Αλλά παρόλα αυτά ακόμα και όταν το κάνουν ο κόσμος μένει χωρίς δουλειά και γι' αυτό τους βοηθάμε να βρούνε κάποια νέα απασχόληση. Η χρηματοδότηση λοιπόν του Ταμείου δεν ωφελεί την επιχείρηση γιατί η επιχείρηση εν μεταξύ έχει απολύσει, έχει φύγει, έχει κλείσει, έχει είπαμε αναλάβει τις υποχρεώσεις της αλλά δεν συμμετέχει πλέον. Λοιπόν αυτά ελπίζω να απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις. Εάν υπάρχουν συμπληρωματικές είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όταν θα ε, λάβουμε τις αποφάσεις για το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης, να μας δώσετε στατιστικές, δηλαδή τα χρήματα σε ποιες χώρες κατευθύνθηκαν και σε ποιους τομείς. Να μάθουμε δηλαδή ποιοι ήταν οι τομείς οι οποίοι επλήγησαν περισσότερο από την παγκοσμιοποίηση. Εγώ μάλιστα θα ήθελα να περιληφθούν και οι αγρότες. Μπορεί να απαντήσει η Επιτροπή. Ναι, εύκολο είναι αυτό. Μπορώ να σας στείλω το ε, link για την ιστοσελίδα μας. Εκεί βάζουμε βεβαίως, ε, ενημερώνουμε την ιστοσελίδα αυτή κάθε εβδομάδα. Ναι, στείλτε το παρακαλώ στη γραμματεία της Επιτροπής ε, Περιφερειακής Ανάπτυξης και εμείς θα το διαβιβάσουμε σε όλους. Κύριε Γκάιερ, θέλετε να μας πείτε κάτι. Ναι. Τι να πω τώρα παραπάνω από αυτά που είπε η εκπρόσωπο τη Κομισιόν. Εγώ είμαι και μέλος της Επιτροπής προπολογισμών. Και αναλαμβάνω και τι ευθύνε μου όταν έρχεται ένα, όταν έχει μια αίτηση μάλλον για χρήματα από το ε, Ταμείο Παγκοσμιοποίηση. Εγώ θεωρώ πάντως το ταμείο αυτό υποχρηματοδοτούμενο. Εάν τώρα ε, πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να στηρίξει και τους Γιωργούς δεν θα μου ήταν ε, τόσο ευχάριστο αυτό. Τώρα, όπως εξήγησε τη διαδικασία η Κομισιόν, Θα αρχίσουν βέβαια, σύμφωνα με αυτά που άκουσα, να αρχίζουν και οι, συνάδελφοι των φιλελευθέρων να διαμαρτύρονται. Τέλος πάντων, δεν πρόκειται το, το ταμείο αυτό να, να συνδεθεί πάρα πολύ στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αυτό είναι σίγουρο. Έχω τώρα τροπολογίες και μέχρι να συμφωνήσουν οι συνάδελφοί μας των άλλων συναρμόδιων επιτροπών θα δούμε, θα έχουμε χρόνο. μπορούμε να προχωρήσουμε και τότε σε ψηφοφορία των προτάσεων. Δεν ανησυχώ λοιπόν. Μπορούμε δηλαδή να ολοκληρώσουμε πρώτα την εργασία μας. Τώρα, για τους αγρότες, μια τελευταία λέξη. Έχω διαφορετική άποψη από τον κύριο Κέλλη, διότι θεωρώ ότι οι αγρότες έχουν χρόνο επαρκή στη διάθεσή τους, σε περίπτωση δηλαδή ε, Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών και γιατί αυτή είναι η αιτιολογία που προβάλλει η Κομισιόν να προσαρμοστούν γιατί τώρα το ε, Ταμείο Παγκοσμιοποίησης να επεκταθεί για να καλύψει και τους αγρότες. Η γεωρική οικονομία έχει τη δυνατότητα να προσαρμοστεί. Προβλέπονται στις συμφωνίες αυτές μεταβατικές περίοδοι και μπορούν να δοθούν τέτοιες μεταβατικές περίοδοι, περίοδοι για να επιτρέψουν την προσαρμογή των ε, αγροτών. Εγώ βέβαια δεν είμαι ειδικό τη αγροτική οικονομία. Γνωρίζω, είμαι, είμαι, είμαι ειδικό στου προπολογισμού και στου ελέγχου προπολογισμού, αλλά γνωρίζω ότι η γεωργική οικονομία έχει ε, στη διάθεσή τη γεωργική πολιτική, αν θέλετε, τα μέσα για να μην αφήσει απροστάτευτους του γεωργούς. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Παγκοσμιοποίησης να μην πάει να γίνει ωστόσο ένα σούπερ μάρκετ όπου όλοι όσοι ε, υφίσταται κάποιες αρνητικές επιπτώσεις, θα ξέρουν ότι μπορούν να πλώσουν το χέρι και να πάρουν. Εάν ωστόσο αυτό βοηθήσει να κερδίσουμε κάποιους ψήφους υπέρ και στο Συμβούλιο, αυτό ίσως είναι θεμητό. Πάντως, το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης δεν είναι και τόσο μεγάλο ώστε να μπορέσει να ικανοποιήσει όλες αυτές τις ανάγκες. Πράγματι θα πρέπει να ρίξουμε το βάρος στην προσπάθεια στήριξης των πλέον ευάλωτων και να σκεφτούμε, διότι αυτό που αναφέρεται στους αυτοαπασχολούμενους οπωσδήποτε περιλαμβάνει και τις μικρές και πάρα πολύ μικρές επιχειρήσεις, τις μικροεπιχειρήσεις. Προτιμώ πάντως ο κύκλος των δικαιούχων να μην διευρυνθεί υπερβολικά, έτσι ώστε τουλάχιστον έχει τη δυνατότητα να δράσει κάπως το τάμιο αυτό. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε την εξή κατάσταση τώρα. Η ημερομηνία α, της ψηφοφορίας στην Επιτροπή Επασχόληση είναι 21η Ιουνίου. Στο μεταξύ έχουμε κάποια νέα στοιχεία. Η Επιτροπή Γεωργίας ζήτησε εφαρμογή του άρθρου 50 θα αποφασίσει η διάσκεψη των Προέδρων Επιτροπών στις 22 Μαΐου στο Στρασβούργο και μετά, μέσω μετά η συνδιάσκεψη των Προέδρων των Ομάδων. Θα δούμε αν θα καθυστερήσει η διαδικασία λόγω επιμερισμένης αρμοδιότητας μεταξύ των δύο επιτροπών. Βέβαια, μπορούμε να το διακινδυνεύσουμε και να θεωρήσουμε ότι θα ικανοποιηθεί το αίτημα της Επιτροπής Γεωργίας για συναρμοδιότητα και θα είναι θετική αντίδραση της διάσκεψης των Πρόεδρων Επιτροπών ως προς το αίτημα της ε, Επιτροπής Άγκρη. Οπότε σήμερα μπορούμε να αποφασίσουμε να καθορίσουμε την προθεσμία για την ε, υποβολή τροπολογιών μια κυρία έτοιμη γνωμοδότηση την 3η Μαΐου. Οπότε εμείς ε, θα ετοιμάσουμε την γνωμοδότησή μας εγκαίρως ό,τι και γίνει ως προς την αρμοδιότητα των Επιτροπών ε, Γεωργίας και Απασχόλησης. Έτσι είμαι εκτό ασφαλού. Εγώ θα προτιμούσα να αποφύγουμε που διακινδυνεύσουμε. Δεν ξέρω τι θα πει ο εισηγητή. Μια και είναι έτοιμη η γραμμαδότηση όμω, λέω να καθορίσουμε τη διορία για τις τροπολογίες την 3η Μαΐου Και αν στο μεταξύ αλλάξει η κατάσταση, θα δούμε αν θα προσαρμόσουμε και εμείς το δικό μας χρονοδιάγραμμα. Δεν ξέρω όμως ποια είναι η γνώμη του συγγετού του κυρίου Γένς Γκάιερ. Εγώ θα ήθελα κάποια στιγμή να εξετάσουμε κατά πόσο θα δικαιωθεί η Επιτροπή Γεωργίας αν συμμετάσχουν σύμφωνα με το άρθρο 50 θα έχουν επί της ουσίας αρμοδιότητα. Για, μα, εμείς δεν, για μας δεν είναι κατεπήγον, έχουμε λοιπόν δυνατότητα να προβλέψουμε κάποιο χρόνο. Οπότε παραλαμβάνω, αν περιμένουμε την απόφαση της διάσκεψης των Προέδρων Επιτροπών για το αν θα ε, ε, κατακυρωθεί συναρμοδιότητα στην Άγκρη θα περιμένουμε. Αν χάσει όμως η Επιτροπή Άγκρη, μάλλον θα αλλάξει το χρονοδιάγραμμά της Επιτροπή Απασχόλησης, δηλαδή η ψηφοφορία στην 21η Ιουνίου. Οπότε θα προλάβουμε εμείς εγκαίρως να καταθέσουμε τη γνωμοδότησή μας. Δεν θα προλάβουμε να μεταφράσουμε τη γνωμοδότηση της τροπολογίας και ούτω καθεξής. Εγώ προτιμώ να είμαστε έτοιμοι για πάνω δεχόμενο και μια και είναι έτοιμη γνωμοδότηση να προσδιορίσουμε το συντομότερο δυνατό την διορία για τις τροπολογίες, αλλά από εσάς εξαρτάται κύριε Σιγητά. Γκάιερ. Αλλιώ το κατάλαβα στην αρχή. Συμφωνώ όμως τώρα με αυτό που είπατε κυρία Καλά, Καλώς, ευχαριστώ. Οπότε, η ημερομηνία για τι τροπολογίε λήγει 3 Μαΐου και αν μέχρι τα τέλη Μαΐου αλλάξει η κατάσταση, θα το ξανασκεφτούμε. Αν χρειαστούν και άλλες αλλαγές, θα δούμε. Αυτό είναι το τελευταίο σημείο της σημερινής, ε, του σημερινού προγράμματος. Η επόμενη μας συνεδρίαση θα γίνει στις 8 Μαΐου, Τρίτη, πρωί και απόγευμα. Μία ημέρα συνεδρίασης πλήρης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους διερμηνείς, λέει Πρόεδρος. Λίγεται η συνεδρίαση.